So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στη συνεδρίασή Μα Είμαστε Δευτέρα απόγευμα και έχουμε και πολλού συναδέλφου παρόντε. Α ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια έχουμε ανακοινώσεις του Προέδρου. Την περασμένη εβδομάδα καταλήξαμε σε συμβιβαστική λύση για τον κανονισμό για τα βιοκτώνα. Πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο. Έχουμε ε, το Σεβέζο 3 και τις συνεχισόμενες ε, διαπραγματεύσεις και Υπάρχει μία αλλαγή στην Επιτροπή μας. Ο Βόλφκαν Klintz δεν είναι πλέον εκπρόσωπος, αλλά ο Ερζέ Κόσελτ είναι ο διάδοχός του. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας καλωσορίζουμε, αγαπητέ συνάδελφε. Έχουμε αρκετές ανακοινώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη έκθεση για την οικονομική κρίση στην Ευρώπη και για τη χρηματοδότηση της προστασίας ε, του κλίματος και ε, υπάρχει ε, κάποιο έλλειμμα στη βοήθεια την οποία μπορούμε να δίνουμε στις χώρες του τρίτου κόσμου και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει όσον αφορά τη συμπληρωματική χρηματοδότηση για το 2012. Υπάρχει άλλη μία μελέτη την οποία έχει κάνει η Επιτροπή σχετικά με ε, την μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο συνεπάγεται τεράστια έξοδα ε, για τον τομέα της υγείας και για άλλους τομείς λόγω της μη εφαρμογής ε, των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ε, η έκθεση για τις ακραίες ε, καιρικέ συνθήκες και το 2011 σε όλες τις υπήρου είδαμε ότι υπήρχαν φυσικές καταστροφές και αύξηση μάλιστα των φυσικών καταστροφών λόγω είτε ξηρασία είτε πλημμυρών και καταιγίδων. Περνάμε τώρα στο βασικό σημείο της σημερινής μας σημερινής διάταξης και εδώ θέλω να καλωσορίσω τον επίτροπό μας, τον Γιάννη Σποτότσνικ, πολύ σημαντικός επίτροπος για τη δική μας επιτροπή. Καλώς ήρθατε κύριε επίτροπε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες από το δικό σας τομέα και σήμερα το θέμα της συζήτησή μας είναι μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και εδώ υπάρχει ο χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι εξαιρετική η σύμπτωση, διότι σήμερα συζητάμε την έκθεσή μας για αυτό το θέμα, την έκθεση του συναδέλφου Γκερμπράντι από την προστασία του κλίματος εδώ και χρόνια έχουμε μάθει ότι χρειαζόμαστε Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και σαφώς ε, συνδέονται όλοι οι πόροι τους οποίους υπερχρησιμοποιούμε και γι' αυτό υπάρχει αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία για την Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Ε, πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία. Εντάσσεται και με τη στρατηγική του 2020 και με το χάρτη πορείας θα έχουμε ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Επίτροπε για να μας παρουσιάσετε τον οδικό χάρτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, μέλη τη Επιτροπής. Ξεκινώ μια κοινοβουλευτική εβδομάδα, γιατί αύριο είμαι στην Επιτροπή Αναφορών, την επόμενη μέρα είμαι στην Επιτροπή Ήτρε. Στην Επιτροπή Αναφορών δεν θα συζητήσουμε βέβαια τα ίδια θέματα. Έχουμε άλλα θέματα, αλλά στην Επιτροπή Ήτρε θα συζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα, την αποτελεσματικότητα των πόρων η αποτελεσματικότητα των πόρων σίγουρα θα είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει βέβαια και την Επιτροπή Αναφορών. Ξεκινώ με το Victor Hugo, με το Victor που είπε ότι ποτέ, τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από μια ιδέα που έχει οριμάσει. Από την ακρόασή μου εδώ πριν από δύο χρόνια, ξέρετε ότι η αποτελεσματικότητα των πόρων πάντοτε κατά την θητεία μου αποτέλεσε προτεραιότητα για μένα και τους τελευταίους μήνες ε, έθεσα ως καθήκον μου το να προωθήσω την αποτελεσματικότητα των πόρων και από τις αντιδράσεις που έχω λάβει από ακαδημαϊκούς κύκλους, από επιχειρηματίες, από υπουργούς, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι σαφές ότι έχει φτάσει πλέον ε, η στιγμή να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα των πόρων είναι αναπόφευκτο το να θέσουμε κάποιους περιορισμούς στη χρήση των πόρων και να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα. Παράλληλα αποτελεί και μια ευκαιρία γιατί θα δώσει ένας μας στην δημιουργικότητα, την καινοτομία και θα καθοδηγήσει νέες πολιτικές, θα δώσει κίνητρα σε επιχειρηματικές αποφάσεις και θα μετασχηματίσει την καθημερινή μας ζωή με γενικότερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Γνωρίζω ότι ε, μιλώ ενώπιόν σας ε, σε ένα ακροατήριο δηλαδή που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα της αποτελεσματικότητας των πόρων και δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να σας πείσω ότι αυτή είναι η σωστή πορεία. Γνωρίζω ότι εσείς ήδη δουλεύετε πάνω σε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, ε, όπου η είναι ο κύριο Γκέρμπεν Γιάνν Γκερμπράντι. Το κοινό μας καθήκον θα είναι να πείσουμε τους υπολείπου μέσα στα θεσμικά μας όργανα, αλλά και εκτός των θεσμικών οργάνων. Πρέπει να τους πείσουμε σχετικά με τα επιχειρήματα και ως προς τη θεωρία και ως προς την πράξη τα οποία χρειαζόμαστε για να μπούμε στο σωστό δρόμο. Θα πρέπει να πείσουμε όλους για το πώς ακριβώς θα μετασχηματίσουμε την πορεία της Ευρώπης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των πόρων. Από το θεωρητικό πώς τώρα πρέπει να περάσουμε στο πρακτικό πώς ε, της αποτελεσματικότητας των πόρων. μετά ε, τον, ε, μετά το ορόσημο των 7 δισεκατομμυρίων που έχει φτάσει πλέον ο πληθυσμός ε, του πλανήτη μας, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι μέχρι το 2050 θα αυξηθούν πάρα πολύ τα ποσοστά κατανάλωση σπόρων κατά 70% μέχρι το 2050 και παράλληλα θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι πόροι που μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούνται με μη διώσιμο ε, τρόπο. Θα χρειαστούμε μέχρι το 2050 τριπλάσιους πόρους αν συνεχίσουμε την πρακτική που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε ε, να αλλάξουμε πορεία, να χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους ή διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την οικονομική μας ανάπτυξη. Και βλέπουμε με την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών ε, ότι είχαμε μια συνεχή πορεία ανάπτυξης των τιμών κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα εκτός των περιόδων πολέμων. Έχει περάσει η εποχή των φθηνών πρώτων υλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία θα επηρεάσει την ε, οικονομική μας και κοινωνική σταθερότητα κατά τις επόμενες δεκαετίες. Είναι σαφές στις περισσότερες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 87% των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν αυξανόμενες τιμές ε, των πρώτων υλών τα επόμενα χρόνια και το κόστος των πρώτων υλών ε, αντιπροσωπεύει το, το κόστος των ε, υλικών αντιπροσωπεύουν το 40% και λιγότερο από 20% αντιπροσωπεύει η εργασία. Αυξάνονται λοιπόν οι τιμές των πρώτων υλών, πράγμα το οποίο ε, σαφώς επηρεάζει ε, την ε, αποδοτικότητα των εταιριών και εδώ πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχουν αγορές οι οποίες να λειτουργούν σωστά όσον αφορά το καθαρό αέρα, το καθαρό νερό ή τα αλλιεύματα ή το οικοσύστημα γενικότερα. Και εμείς έχουμε το καθήκον να διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύουμε προστατεύονται οι ευπαθείς πόροι, ούτως ώστε να προετοιμάζονται οι πολίτες αλλά και η βιομηχανία για τα μελλοντικά βήματα. Πρέπει να αποσυνδέσουμε ε, τους ε, πόρους από την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να δώσουμε σαφή μηνύματα προς τις επιχειρήσεις και προς τους καταναλωτές και να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη τους και την προβλεψιμότητα ώστε να μπορούν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής και πολιτικής που θα ακολουθήσουν. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια τα οποία κλειδώνουν τις οικονομίες μας, τις κοινωνίες μας και τους πολίτες μας στο τωρινό σύστημα. Πώς μπορούμε ε, να διευρύνουμε τους ορίζοντες στη λήψη αποφάσεων. Πώς μπορούμε να επιφέρουμε τις σημαντικές καινοτομίες που απαιτούνται σε πολλούς τομείς. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ζήτηση για πράσινα προϊόντα, οικολογικά προϊόντα σε πολλούς τομείς στον οδικό χάρτη ακριβώς αυτό το πώς προσπαθούμε να απαντήσουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε στην αποτελεσματικότητα των πόρων στην Ευρώπη. Για μένα αποτελεί προτεραιότητα αυτό το θέμα. Και καταρχήν θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι δικός μου χάρτης πορείας, είναι χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πόρων. Εγκρίθηκε από όλο το σώμα των επιτρόπων. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινό όραμα για το τι χρειαζόμαστε για το 2050 και για την πορεία μας μέχρι τότε για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί ως ηγέτες εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η αποτελεσματικότητα των πόρων αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία στα πλαίσια της ατζέντα του 2020 και για το περιβάλλον αλλά και για την ανταγωνιστικότητα, για την αηφόρο ανάπτυξη. Πάνω σε αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία λοιπόν ταιριάζει και αυτός ο δικός χάρτης ούτως ώστε να έχουμε συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το όραμά μας και θα ήθελα να σας το επαναλάβω. Μέχρι το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει αυξηθεί κατά τρόπο ώστε να σέβεται τους περιορισμούς που υπάρχουν για τους σπόρους και τις δυνατότητες του πλανήτη μας. Η, οικονομία μας θα παραμένει ανταγωνιστική και πολυσυλλεκτική και θα προσπαθεί να έχει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος. Θα γίνεται συνετή διαχείριση των πόρων, θα πρέπει να έχουμε επιτύχει σημαντικά ορόσημα όσον αφορά την προστασία του κλίματος, να προστατεύουμε τα οικοσυστήματα και να τα έχουμε αποκαταστήσει κατά τρόπο βιώσιμο. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά και ο δικός χάρτης θέτει κάποια ορόσημα μέχρι το 2020. Έχουμε τονίσει τρία ε, σημεία, τρει τομεί τη ζωή μα. τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τα τρόφιμα και τι μεταφορέ. αυτά τα τρία σημεία, αυτοί οι τρει τομεί αποτελούν περίπου το 80% ε, των ε, επιπτώσεων των ανθρώπων επί των πόρων μας από την νομοθεσία για τα απόβλητα μέχρι την νομοθεσία για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού και θα πρέπει να ληφθούν σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις ταυτόχρονα. Όλα αυτά εντάσσονται για πρώτη φορά στο ευρύτερο πεδίο του διαρθρωτικού μας οικονομικού προγράμματος. Ο δικός χάρτης θέτει ορόσημα για το 2020, κατευθύνσεις πολιτικής και προτεραιότητες. Βέβαια δεν ορίζει λεπτομέρειες τις 24 σελίδες που περιλαμβάνει, δεν μιλά για κάθε νέα πρωτοβουλία, για κάθε νέο νομοθετικό κείμενο. Παραδείγματο χάρη ζητούμε ε, περιορισμό των χωματερών μέχρι το 2020, μείωση των ε, επιδοτήσεων, μετακίνηση από φορολόγηση της εργασίας σε φορολόγηση της ε, ρήπανσης του περιβάλλοντος. Για πρώτη φορά προτείνονται μέτρα για τη βιώσιμη γεωργία και για τη χρήση γης ζητείται κινητοποίηση εργαλείων που θα βασίζονται στην αγορά. Ιδίω η στρατηγική έξι για τη διόρθωση των αστοχιών της αγοράς και για τον ε, σωστό καθορισμό των τιμών, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν ε, το πραγματικό κόστος των πόρων και να καθοδηγούν ε, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές προς τη σωστή κατεύθυνση. Νέε πολιτικές που θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις τιμές των πόρων που δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς στην αγορά, όπως είναι η βιοπικιλότητα, η ποιότητα του ύδατος και του ατμοσφαιρικού αέρα. Ο οδικός χάρτης προτείνει η φορολογία να μεταθέσει το βάρος της στη ρήπανση και στους πόρους, και να μην χρησιμοποιούνται ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ταυτόχρονα και φορολογική ε, πολιτική ε, προσαρμοσμένη και θα χρησιμοποιούνται οι πόροι με αποτελεσματικό τρόπο. Εντάξει. Για να αποφύγουμε δυσμενείς επιπτώσεις χρειαζόμαστε ε, μέσα και από την πλευρά της προσφοράς και από την πλευρά της ζήτησης. Από την πλευρά της προσφοράς ε, θα πρέπει να διευρύνουμε παραδείγματος χάρη τα κριτήρια για τον οικολογικό σχεδιασμό. Και στην, από την πλευρά της προσφοράς, θα ε, από την πλευρά της ζήτησης θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια αγορά βιώσιμων προϊόντων που παράγονται με αηφόρο τρόπο, βελτιώνοντας παραδείγματος χάρη την πολιτική μας στον τομέα των κριτηρίων για τις οικολογικές συμβάσεις. Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις και στις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από την διαδικασία αυτή. Δεν έχουμε βέβαια επιτύχει ακόμη αυτό το στόχο και γι' αυτό ο δικός χάρτης προτείνει να ξεκινήσουμε με ένα δίκτυο που θα είναι η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα των πόρων και στη συνέχεια ε, να προχωρήσουμε με δείκτες για τα υλικά, για τον άνθρακα, για το και για τη γη. Παράλληλα, έχουμε ορίσει κάποιους συγκεκριμένους δείκτες για συγκεκριμένες πολιτικές και αυτό θα βελτιώσει τους στόχους που έχουμε ιδίως στον τομέα των αποβλήτων. Αυτά μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Βέβαια δεν θα σταματήσουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Με τον οδικό χάρτη ε, ξεκινάει μια διαδικασία πολλών σταδίων με πολλούς εμπλεκομένους ε, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να ορίσουμε συνεκτικούς στόχους και δείκτες όταν υπάρχει μια κρίση θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε κάτι καλύτερο. Η τωρινή κρίση, όσο δύσκολη και αν είναι, δίνει ευκαιρίες για μεταρρυθμίσεις πολιτικών, τόσο ώστε να διασφαλίσουμε ε, μια μελλοντική πορεία προς ε, την επιτυχία. Και η αποτελεσματικότητα των πόρων θα είναι κάτι το οποίο θα ενταχθεί πλήρως στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν την αποτελεσματικότητα των πόρων εγγενές τμήμα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Κάποια πρώτα βήματα είναι το να ε, μην υπάρχουν ουσίες οι οποίες είναι επιβλαβείς προς το περιβάλλον και η φορολογία να μετακινηθεί ε, από τη φορολόγηση της εργασίας στη φορολόγηση της ρήπανσης θα πρέπει να δώσουμε μέσω της καινοτομίας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες αγορές ε, για τις πρώτες και θα πρέπει οι δημόσιες αρχές ε, να ε, φροντίσουν οι δαπάνες τους να γίνονται με τρόπο οικολογικά σωστό. Θέλουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα Life Sin και Παράλληλα, οι πρώτες ε, προτάσεις της Επιτροπής για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα ακολουθήσουν μια οικολογική ε, προοπτική. Ευχαρίστω να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η υποστήριξή σας θα είναι πολύτιμη σε αυτό το πλαίσιο, ούτως ώστε και ο προϋπολογισμός μας να διέπεται από οικολογικές αρχές. Κυρίε και κύριοι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και βασίζομαι στην υποστήριξή σας, ιδιαίτερα για τις συγκεκριμένε προτάσεις, οι οποίες ε, θα φτάσουν κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω την αρχή μιας ιστορίας. Τον περασμένο μήνα η εφημερίδα Guardian ζήτησε από τους αναγνώστες να στείλουν μια επιστολή στο μωρό που γεννήθηκε ως υπαριθμόν 7 δισεκατομμυριωστός πολίτης ε, του πλανήτη μας. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτό το παιδάκι. Καλώς ήρθε σε αυτή την κατάσταση κρίσης, όπου εμείς έχουμε φροντίσει ο πλανήτης μας να υπερθερμαίνεται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά η δική σου γενιά μπορεί να είναι η γενιά η οποία είτε θα καταστρέψει τον πλανήτη, είτε θα τον σώσει. Θα πρέπει να βρείτε τι λένε οι επιστήμονες και να κάνετε κάτι να βοηθήσετε έστω και με μικρά βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, πολύ ωραία. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Γιάννη Ποτότσνικ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενημερωτική εισήγησή σας γιατί χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με ε, επαρκή οικονομικούς πόρους. Ξεκινήσατε από τον Βίκτορ Ουγκό και φτάσατε μέχρι το μωρό αυτό το, που είναι ο 700 έβδομος δισεκατομμυριωστός πολίτης του πλανήτη. Μέσα από όλα αυτά εκφράσατε τις ανησυχίες σας για τον πλανήτη. Πράγματι, αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται εδώ για τον οδικό χαρτί του συλλόγου, του συνόλου των επιτρόπων και όχι του ε, επιτρόπου περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν ένα θέμα που είναι δεσμευτικό και για άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι επίση σαφέ ότι εφόσον μιλάμε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο των επόμενων ετών, πρέπει να εξευρεθούν οικονομικοί πόροι έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει το μέλλον τη. Ε, θεωρώ ότι το θέμα αυτό πρέπει να γίνει η βάση όλων των σεμιναρίων που θα ακολουθήσουν, ε, βάσει αυτού να κρίνουμε αν βελτιωνόμεθα ή όχι. Εμένα ε, με ενδιαφέρει το κατά πόσον το έβδομο πρόγραμμα δράσης για την επόμενη χρονιά, κατά πόσον το πρόγραμμα αυτό έχει σχέση με τον χάρτη πορείας και με άλλες ε, λεπτομέρειες που έχουμε σκεφτεί μέχρι το 2020. Για το θέμα αυτό υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε λοιπόν με τους ε, συντονιστές. Ο πρώτος εισηγητής σε τρία λεπτά. Ο κύριος Σίμπα. Ε, εσείς ο πρόεδρος, εσείς εκείνος ε, που κατανέμεις το χρόνο και βεβαίω είναι δικό καθήκον να κατανέμεις το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την εισηγησή σας. Ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Μετά λοιπόν από την ανάλυση που ακούσαμε και που σε μεγάλο βαθμό συμμεριζόμαστε, ε, αν και βέβαια ε, αυτό ε, το απεσιόδοξο στοιχείο που αποδώσατε, εμένα δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική περιβάλλοντος πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και μόνο με την αισιοδοξία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα σωστά πολιτικά εργαλεία. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, αυτή η στρατηγική για την ε, Ευρώπη ε, ικανοποιητικών πόρων έχει εγκριθεί από το σύνολο των επιτρόπων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω το εξής. Εφόσον πρόκειται για το περιβάλλον και εφόσον ε, το θέμα αυτό περιλαμβάνει πολλές προεπτάξεις, γιατί δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο που έχετε στα χέρια σας, τον κανονισμό. Σε τελική ανάλυση διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές οδηγίες, πολλοί κανόνες. Τα κράτη-μέλη όμως ε, υπολείπονται κατά πολύ του αναμενόμενου, ε, κυρίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το θέμα των αποβλήτων. Ε, στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές και διαφορετικές νομοθεσίες. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ελέγξει περισσότερο την εφαρμογή των κανόνων. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αυτά επί των οποίων έχουν συμφωνήσει. Και εφόσον δεν το πράττουν, η Κομισιόν επεμβαίνει και μάλιστα με σκληρά μέτρα. Ο κανονισμός λοιπόν είναι ένα πολύ απλό εργαλείο ε, που προσφέρει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να κάνει όλα αυτά, ε, να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν την συμφωνημένη πολιτική, πράγμα που δεν επιτρέπει η οδηγία. Νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ε, πρέπει ακόμα να κάνουμε πάρα πολλά. Κατά τα άλλα, περιμένουμε ακόμα αυτή την οδηγία για τα βιοαπόβλητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λιγάκι αποκλίνουσα άποψη από εμάς. Νομίζω όμως ότι το θέμα αυτό τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, χαιρετίζω αυτά που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρασίνισμα της ε, περιφερειακής και της γεωργικής πολιτικής. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι σε τελική ανάλυση τι θα απομείνει. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις που είναι επιβλαβή ζημιογόνες για το περιβάλλον, αυτές ε, θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή θα καταργηθούν. Αναφέρομαι κυρίως στον τομέα των υδάτων. Αν δείτε λιγάκι την ε, Γεωργία, εκεί το νερό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ελπίζω ε, να καταλήξουμε σε μια λύση, να μην υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα σε χώρες με έντονη λειψιδρία. Όσον αφορά το περίφημο blueprint, είσαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα. Ε, και θα μπορέσουμε και εμείς νομίζω να συνεισφέρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που από ό,τι φαίνεται σε αυτόν τον τομέα έχουμε βρει το σωστό εργαλείο. Για άλλη μια φορά λοιπόν από δική μας πλευρά σας εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας και θα θέλαμε να σε ενθαρρύνουμε να ε, επιπλήξετε τουλάχιστον να επιπλήξετε τα κράτη-μέλη αν δεν εφαρμόζουν αυτά επί των οποίων έχουν συμφωνήσει. Η Λίντα Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προτάσεις σας και νομίζω ότι οι πιο πολλοί συνάδελφοι εδώ θα συμφωνήσουν μαζί μου. Εμείς είμαστε η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε το μήνυμα αυτό να το βοηθήσουμε να διαδοθεί Έχουμε εδώ τον κύριο Φλόρο, ο οποίος μπορεί να μας ε, πει τι γίνεται με τι διαπραγματεύσει που γίνονται στο θέμα ε, με το Συμβούλιο. Ε, βλέπω ότι γνέφει. Εμείς θα νομοθετήσουμε για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, ξέρουμε ότι έχετε δίκιο σε αυτά που περιγράφετε και θεωρώ πω και η απόκριση του Συμβουλίου δεν θα είναι ικανοποιητική. Ε, τώρα για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, για την κοινή γεωργική πολιτική και για την αλληλεία, δεν ξέρω αν εσείς συνεργάζεστε με τις άλλες γενικές διευθύνσεις. Δεν ξέρω αν θα εξασφαλίσετε πως το θέμα της αλληλείας και της γεωργίας κάτι θα αλλάξει. Γιατί για να μην ειλικρινής, αυτό το οποίο ακούω στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι προσπαθούν να καθυστερήσουν στους διαδρόμους μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πόσο δραστήριοι είστε στη συζήτηση των θεμάτων αυτών και με τις άλλες αρμόδιες επιτροπές αλλά και με το Συμβούλιο. Αναφερθήκατε σε αυτό το μωρό και διάβασα στους Financial Times ότι σήμερα περιμένουν ε, μία έκρηξη σε άλλες ε, πηγές ενέργειας όπως για παράδειγμα οι πίσες, ε, τα τα σχιστολιθικά καύσιμα. Λοιπόν, πείτε μου, εκεί περιμένετε κάποιες εξελίξεις? Γιατί αυτό που ανησυχώ εγώ είναι πως ε, στο μωρό αυτό θα πρέπει να πούμε πως εμείς μάθαμε πολλά αλλά δεν κάναμε τίποτα γιατί δεν μας βόλευε. Και μια τελευταία ερώτηση, την οποία ενδεχομένω δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε σήμερα, είναι για ένα χημικό που ονομάζεται και TCI και TCE, το έχω δει να γράφεται και με τους δύο τρόπους. Η τριο ε, φθοροεθυλίνη που χρησιμοποιείται στους διαλύτες. Έγινε μια μεγάλη μελέτη στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε ε, που τη συνδέουν με την ασθένεια του Πάρκινσον και είναι μια χημική ουσία η οποία αυτή τη στιγμή έχει μπει στη διαδικασία του REACH Οπότε φαντάζομαι πως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον κατάλογο αδειοδότησης. Ε, έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από το φαρμακευτικό λόμπι και από την βιομηχανία να μην μπει η ουσία αυτή στον κατάλογο των ουσιών που χρειάζεται αδειοδότηση. Ελπίζω εδώ να παρακολουθήσετε το θέμα και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες ε, παραπάνω εάν θεωρείτε πως σας ενδιαφέρει τριφθοροεθελήνη. Λοιπόν, είναι αρκετά εύκολο, λέει ο πρόεδρος. Για να περάσουμε λοιπόν και να δούμε αν μπορώ να δώσω τη θέση μου στον κύριο Γκεμπράντη για να πάρει το λόγο πρώτος. Σας ευχαριστώ. <laughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είδατε εμείς είμαστε πολύ ε, αποτελεσματικοί στον χρόνο που κατανέμουμε το χρόνο μας. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω τα όσα είπε η συνάδελφος. Είμαστε η Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος και θα συμφωνήσουμε με τις προτάσεις που έγινε για την αποδοτικότητα, που έγινε για την αποδοτικότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι ίσως εδώ θα έπρεπε να είναι και η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων η οποία θα έπρεπε να στηρίξει τις προτάσεις αυτές για να είμαστε στο 100% των δυνάμεών μας. Αν εξετάσετε τα αριθμητικά στοιχεία που μας έδωσε μόλις ο Επίτροπος, νομίζω πως ε, και σε οικονομικό επίπεδο ήταν πιο λογικό να είμαστε πιο αποδοτικοί στη χρήση των πόρων που έχουμε. Στο έγγραφο εργασία που καταθέτω έχω δώσει και εγώ κάποια αριθμητικά στοιχεία και με εντυπωσιάζει και δεν μπορώ να το πιστέψω πως για, ε, ακόμα και για απλά οικονομικούς λόγους δεν έχουμε αποφασίσει να γίνουμε πιο, να περιορίσουμε τη χρήση των ε, πόρων αυτών. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης η οποία φαίνεται να σφίγγει κάθε μέρα πιο πολύ. Αν διαβάσει κανείς τις ε, εφημερίδες, κάτι τέτοιο θα διαπιστώσει. Είμαι λοιπόν πεπισμένος πως ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξεπεράσουμε με επενδύσεις αυτή την οικονομική δυστοκία είναι ε, με μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην χρήση των ορυνογιακών πόρων, δηλαδή η βιωσιμότητα και μιλάμε για μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία θα είναι πιο βιώσιμη και πιο αποδοτική στη χρήση των πόρων, θα είναι σε θέση να ξεπεράσει τις σημερινέ οικονομικέ δυσκολίες και να γίνει και πιο ανταγωνιστική. Ρωτώ λοιπόν τον Επίτροπο και ξέρω που συμφωνείτε με τις παρατηρήσεις μας. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως οι συνάδελφοί σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζουν τις προτάσεις αυτές. Γιατί οι φήμες λένε πως ο δικός χάρτης μάλλον θα αναβληθεί. Επειδή ακριβώς διασχίσουμε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβεί. Θα έπρεπε να έχουμε επιταχύνει στις διαδικασίες αυτές έτσι ώστε να κατατεθεί ο δικός χάρτης ακριβώς λόγω της χρονικής συγκυρίας που διανύουμε. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πόσο, σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει και στηρίζει, και αναφέρουμε και βέβαια και σε κάποια κράτη-μέλη, ε, την οικονομική αναγκαιότητα του να γίνουμε πιο αποδοτικοί στη χρήση των πόρων. Ναι. Λοιπόν, 26 επιτροποί, πόσο, πόσο βαθιά πιστεύουν σε αυτό. Νομίζω πως αυτό θέλουμε να ακούσουμε από εσάς. Θα προσπαθήσω και εγώ να μιλήσω αγγλικά. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο και με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσα πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ε, ό,τι μπορεί για να προωθήσει το θέμα αυτό και για να έχουμε μια πιο χρηστή χρήση των πόρων μας. Και μάλιστα νομίζω αυτή η εβδομάδα είναι η, Διεθνής Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα τρόφιμα θα, αύριο θα ψηφίσουμε, την, θα παρουσιάσουμε ένα ψήφισμα για την αποτελεσματικότητα της διατροφικής αλυσίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ε, αν αυτό αληθεύει θα είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία γιατί μπορεί με πολύ ωραίο χρόνο, με πολύ ωραίο τρόπο να κάνουμε ε, καταρχήν είτε ανακύκλωση σε βιοκαύσιμα των ε, απολύτων τροφίμων που έχουμε, είτε να χρησιμοποιούνται εκ νέου με διαφορετική μορφή. Έχουμε αρκετά μεγάλο νομοθετικό έργο και πολλή νομοθεσία η οποία δεν πιστεύω πως χρειάζεται να αυξηθεί γιατί δεν νομίζω ότι τα έγγραφα θα βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Νομίζω θα πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας, να συστήσουμε με τους ε, συμπολίτες μας ε, για την υπευθυνότητα με την οποία θα διαχειριστούμε τους διάφορους πόρους. Δεν ξέρω. Δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα μόνο ε, να ασχοληθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να ε, το αναλάβουν και οι τοπικές κοινωνίες. Λυπάμαι. Μιλάμε, λυπάμαι για τον κακό ήχο ε, στην, στην αίθουσα αυτή, αλλά δυστυχώς οι τεχνικοί δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο Ποτότσου που μας εξέθεσε τις θέσεις του για την αποδοτικότητα των πόρων. Όπως και εσείς χαιρετίζετε αυτή την, αυτό το χάρτη πορείας, έτσι και εμείς αυτήν την αίθουσα είμαστε προς, κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση. Το θέμα είναι πώς θα πείσουμε τις άλλες γενικές διευθύνσεις και πώς θα το προωθήσουμε μέσα στην υφιστάμενη νομοθεσία των κρατών μελών. Επίσης είπατε ότι και οι δείκτες θέλετε να γίνουν τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να μπορέσουν όλα αυτά να συνεισφέρουν προς το κοινό θεματολόγιο της Ευρώπης. Γνωρίζουμε ότι προσπαθείτε να επεξεργαστείτε και τις θέσεις των άλλων γενικών διευθύνσεων και θα ήθελα να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, ε, δηλαδή, ε, σε τι βαθμό νομίζετε ότι αυτοί οι δείκτες θα μπουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, γιατί τότε θα είναι στο βασικό τμήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Οι δείκτε αυτοί πρέπει να ενσωματωθούν σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσω του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα τη φορολογία. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε σε γενικέ γραμμέ για τη φορολογία, όλοι συμφωνούν να μετακινηθούμε από τη φορολογία τη εργασία, τη φορολογία τη χρήση πόρων, αλλά όταν περνάμε σε πραγματικέ πολιτικέ δεν ακούμε πια τα ίδια θετικά λόγια. Θα μπορούσαμε να έχουμε δεχομένως μια οδηγία για την φορολόγηση των πόρων που να αναφέρει σαφώς ότι μετατίθεται η φορολογία από τη φορολογία της εργασίας στη φορολογία των πόρων. Τρίτον, για την βιομάζα. Ε, είναι ένας από τους πόρους στους οποίους υπάρχει σπάνης και ξέρουμε ότι υπάρχει μια πολιτική, υπάρχουν πολιτικές για την ε, βιομάζα και η χρήση της βιομάζας στο ενεργειακό μας σύστημα γνωρίζουμε ότι δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος χρήσης βιομάζας. Αφού τη χρησιμοποιούμε σε διάφορα στάδια, στο τελικό στάδιο μπορούμε ε, να φτάσουμε στην καύση, αλλά μέχρι την καύση πρέπει να έχουμε χρησιμοποιήσει τη βιομάζα αποτελεσματικά. Ξέρω ότι μέχρι το τέλος του έτους υπάρχουν υποσχέσεις για κριτή κριτήρια βιωσιμότητας ε, για, την, ε, ε, για για τα στερεά υλικά βιομάζα, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδο και αυτό μου δημιουργεί πολλέ αμφιβολίε. σω οι προτάσει δηλαδή να έχουν σχέση περισσότερο με τη δημιουργία ενέα αγορά και να μην είναι τόσο φιλόδοξε ώστε να θέτουν όντω κριτήρια βιωσιμότητα για τη βιομάζα. Γιατί όταν συζητάμε τα θέματα αποτελεσματικότητας των πόρων είναι απαραίτητα τα κριτήρια για τη βιομάζα. Μέχρι τα τέλη του έτους λοιπόν τι μπορούμε να προσδοκούμε. Καλύτερα να έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση και καλές προτάσεις παρά να έχουμε κάποιες προτάσεις που απλώς θα επιδεινώσουν την κατάσταση για τη χρήση βιομάζας. Ευχαριστώ πολύ ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Καλωσορίζω το έγγραφο που μας παρουσιάσατε με τον οδικό χάρτη. Αλλά κάπως απογοητεύτηκα διότι αυτό το έγγραφο είναι αρκετά ε, γενικό και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα και απογοητεύομαι κάπως ε, διότι μιλώ με εκπροσώπους της βιομηχανίας στην Ευρώπη και μου λένε ότι ε, μιλάτε μεν για το σύστημα, αλλά τι κάνετε στην πραγματικότητα. Και ποια νομίζετε ότι είναι τα πραγματικά βήματα τα οποία μπορεί πραγματικά η βιομηχανία να προωθήσει. Όταν φτάνουμε σε τέτοια πρακτικά θέματα δεν υπάρχει καμία απάντηση. Ε, και εδώ έχω λάβει ένα έγγραφο που το έχω μπροστά μου από ένα γνωστό σύνδεσμο ε, ε, επαγγελματικό και διαβάζοντάς το βλέπω ότι οι συμβουλές είναι πολύ λίγες για την πρακτική πρόοδο. Τέλος πάντων, εσείς κύριε Επίτροπε, αν έχετε πολιτική υποστήριξη, γιατί και στην Επιτροπή μας πολύ συχνά δεν έχουμε τέτοια υποστήριξη. Πολλοί συνάδελφοι παίρνουν το λόγο αλλά δεν έχουν πύχηση στις χώρες τους στα αντίστοιχα ε, υπουργεία. Ε, στον τομέα των αποβλήτων, παραδείγματος χάρη, ε, θα πρέπει πολλοί από τους συναδέλφους να απευθυνθούν στις πρωτεύουσές τους και να προσπαθήσουν να πείσουν εκεί τους αρμοδίους ε, να υποστηρίξουν τις προτάσεις της Επιτροπής. Ελπίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή θα έχει μεγαλύτερη υποστήριξη όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα. Να φανεί ότι οι Βρυξέλλες έχουν κάποια επιρροή και στο Παρίσι και στη Ρώμη και στις, ε, στην κάθε πρωτεύουσα. Με ενδιαφέρει να δω πού βρίσκεται η υλοποίηση όλων αυτών. Και ο συνάδελφο Ρίχαρτ Ζέμπερ είπε ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε περισσότερο θετικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ σε αυτή την αίθουσα δέκα φορές ζήτησα τους διευθυντές της Γενικής ε, Διάθεσης Περιβάλλοντος ε, τι γίνεται με την υλοποίηση και πάντοτε την ίδια απάντηση μου δίνουν ότι υπάρχει μια έκθεση και η έκθεση αυτή ε, μας αναγγέλει τις τραγικές συνέπειες αλλά θα ήθελα από αυτούς που βρίσκονται στην ηγεσία να δω ότι πραγματικά εμπλέκονται και πραγματικά υποστηρίζουν αυτές ε, τις ε, προτάσεις και ενοιολογικά και στην πράξη. και ξέρουμε και οι συνάδελφοι το είπαν πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να περάσουμε σε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε μπορούν ε, ε, να αλλάξουν ε, οι συνθήκες για τα απόβλητα, παραδείγματο χάρη, να αλλάξουν οι προτεραιότητες που τίθενται για τις χωματερές, να αλλάξουν οι νομοθεσίες για την κάθιση των αποβλήτων, να βελτιωθεί η κατάσταση για τα απόβλητα και στην Ανατολική, στις χώρες της σχετικής και Ανατολικής Ευρώπης η έκθεση με βρίσκει σύμφωνα θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε περαιτέρω. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ξέρω ότι όλοι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας ε, ε, είναι πεπισμένοι και πραγματικά πιστεύουν και στη Βρυξέλλες και στη χώρα τους αυτά τα οποία υπερασπίζονται εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγησή σας και την φιλόδοξη έκθεση που συντάξατε ε, και εμεί ε, θα σας στηρίξουμε. Μπορείτε να απολογίσετε σε αυτό γιατί και εμείς είμαστε φιλόδοξοι και ίσως και πιο φιλόδοξοι από εσάς. Πρόκειται λοιπόν για μια θαυμάσια ιδέα. Αυτή η έκθεση να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι χώρες, ε, τα κρατη να αναφέρονται ως προς την πρόοδο που επιτυγχάνεται. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η ανακύκλωση και για την ανακύκλωση θα υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή ε, θα μας υποβάλλετε κάθε χρόνο εκθέσεις ε, σε σχέση με την ανακύκλωση. Γιατί υπάρχουν εκθέσεις ε, για τα απόβλητα, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε για τους στόχους αν θα υπάρχει το ίδιο. Και όσον αφορά τους στόχους, θέλω να ρωτήσω κατά πόσον μιλάτε για την χρήση της γης, γενικά για τη χρήση, αυτό σχετίζεται με στόχους. Και θα ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, κύριο Φλόρενς, που μόλις τώρα μας είπε ότι θέλουμε να σας στηρίξουμε όσον αφορά την απαγόρευση χωματερών. Εμείς το έχουμε ζητήσει αυτό, υπάρχει απαγόρευση ανοιχτών χώρων ταφής και ε, θεωρώ ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα προχωρήσετε εσείς στή κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, ε, η απαγόρευση ανοιχτών χώρων ε, ταφής. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί επίσης μας ενδιαφέρει ότι δεν θέλουμε να υπάρχει εξαγωγή ε, ηλεκτρονικών και άλλων στοιχείων. Δεν θέλουμε να υπάρχει το WEEE, e e, η οδηγία η σχετική. Αυτό λοιπόν στη τελική ανάλυση τι σημαίνει, ότι θα ζητήσετε μεγαλύτερη ευθύνη των παραγωγών και κάτι άλλο. Εσείς αναφερθήκατε στην ιεράρχηση. Έχουμε συζητήσει για την ιεράρχηση στα βιοαπόβλητα, αλλά γενικά αυτή η ιεράρχηση μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλουμε να γνωρίζουμε τα προϊόντα. Ε, πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σχέση με την προστιθέμενη αξία. Δεν μιλάω για μια υποχρεωτική ιεράρχηση, αλλά τουλάχιστον Θέλουμε να μελετήσουμε το θέμα και να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις. Και τέλος, κάτι άλλο θέλω να πω. Θέλουμε να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσετε στη φορολόγηση των πόρων, γιατί επιθυμούμε επίσης ε, να υπάρχει και μία ε, μακροπρόθεσμη, μία βιώσιμη φορολογική βάση. Θα θέλαμε τις απόψεις από αυτού. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Κοιτάξτε, αυτή τη βδομάδα θα πάμε στην Καλαβρία υπό την προεδρία του κυρίου Πυρίλιο για να δούμε και επιτόπου τι γίνεται με την εφαρμογή τη οδηγία περί αποβλήτων. Και θα γυρίσουμε και θα σα καταθέσουμε τη σχετική έκθεση. Νομίζω και εσεί, κύριε Επίτροπε επισκεφθήκατε την Καλαβρία. Έτσι δεν είναι. Ο κ. Σαρσένη, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι σε αυτή την Επιτροπή και αληθεύει πως Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε και πιο επικριτικά σε αυτά που είπατε, γιατί καλό είναι να πιέζει κανείς τους φίλους του έτσι ώστε να προχωρήσουν. Πιστεύω, ναι, πως αυτό το μωρό που γεννήθηκε, που είναι ο πολίτης που έφερε τον πληθυσμό της γης στα 7 δισεκατομμύρια, δεν θα προλάβει να δράσει. Γιατί δεν θα δώσουμε εμείς περιθώριο χρόνο για να δράσει. Εάν δεν δράσουμε εμείς, τουλάχιστον για την κλιματική αλλαγή, θα είναι πολύ αργά. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξω το θέμα της βιοπικιλότητας. Στην Αγκόγια αναλάβαμε τη δέσμευση ε, να, ότι θα προστατεύσουμε το 70% της... Ε, χερσαίας επιφάνειας. Αν λοιπόν έστω και ονομαστικά σεβαστούμε αυτό το, το όριο, τότε αυτό το 70% μόνο το 70% αυτού το 70% θα προστατευτεί. Μιλήσαμε για, για διπλασιασμό των αξιολογήσεων που γίνονται στα οικοσυστήματα και 50% για τα ζωικά είδη. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια βελτίωση. Δηλαδή θα διπλασιάσουμε ε, ε, τα είδη στα οποία ε, δίδεται αυτή η, πιο προστατευμένη, ο πιο προστατευμένος χαρτισμός, αλλά και πάλι ε, μόνο το 35% των ζωικών ειδών και το 34% των οικοσυστημάτων θα προστατευθούν. Are you planning to take... Thank Πείτε μου λοιπόν, με τι άλλα μέτρα θα πλαισιώσετε αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πάντα όταν έχουμε επισκέπτες και σήμερα έχουμε ε, μια μεγάλη ομάδα τη συναδέλφου Σοφίου Κονή από τη Γαλλία. Σας καλωσορίζουμε θερμά και από την Λατσάνα Σάμπο από τη Ρουμανία και αυτή έχει επισκέπτε και εσείς καλώς ήρθατε και έχουμε και 16 εκπαιδευόμενους στη μετάφραση τη γραπτή μετάφραση που παρακολουθούν και αυτοί ε, το τι συζητάμε. Και σας σας καλωσορίζουμε. Τώρα, επόμενος που θα λάβει το λόγο είναι ο Αλόης Πέιταρλε. Ε, Σπομίναμε na zaslišanjih govorila o potrebi po spremembi paradigme. E, zanima me ocena gospoda komisarja. Δυστυχώς δεν μπορείτε να μιλήσετε σλοβενικά. Ο Επίτροπος σας καταλαβαίνει, αλλά δεν σας καταλαβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που είπατε πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά κανείς δεν το κατάλαβε. Έχουμε σλοβενικά, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, δεν προβλέπονται ε, σλοβενικά σήμερα. Σλοβενικά δεν προβλέπονται ως γλώσσα διερμηνίας για αυτή τη συνεδρίαση. Ξέρω ότι μπορείτε να μιλήσετε και σε άλλη γλώσσα, ότι είστε ευέλικτος άνθρωπος. Έτσι είναι η μελισσοκόμη. Πριν από δύο χρόνια, αρκετοί υποψήφιοι επίτροποι είχαν, είχαν σχολιάσει την ανάγκη του να αλλάξουμε τα μοντέλα που ακολουθούμε. Η ερώτηση μου είναι η εξής λοιπόν. Πού βρισκόμαστε με αυτή την αλλαγή μοντέλου μετά από δύο χρόνια θητείας της Νέας Επιτροπής. Και βεβαίως Πιστεύετε πως η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επηρεάσει την ε, πρόθεση μας αυτή να αλλάξουμε τα μοντέλα που ακολουθούμε, γιατί συνήθως μπορεί να συμβεί ένα από τα εξή δύο. Είτε σε μια εποχή κρίσης να προσπαθήσουν όλοι να κάνουν μια να κάνουν μια προέκταση των όσων ήδη υφίστανται και να χρησιμοποιήσουν τα παλιά μοντέλα αλλά υπάρχει το εξή σενάριο, όταν η κρίση είναι πραγματικά βαθιά, να βρεθούν κάποιες νέες λύσεις που θα αλλάξουν ε, τις συνηθίες μας. Πού ζούμε, τι τρώμε, πώς μετακινούμαστε. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνουμε και θα ήθελα να πείτε εδώ έχουμε αλλάξει μοντέλα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Λόγω του είπε πως οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να ασχοληθούν με μεγαλύτερη, να σταθούν με μεγαλύτερη προσοχή πάνω από τα θέματα αυτά. Δηλαδή τη χρήση των διαφόρων ενεργειακών πόρων με πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας. Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνουν μόνο οι πολιτικοί ηγέτες. Νομίζω ότι όσοι ε, συμμετέχουν στην προετοιμασία αυτής της απόφασης θα πρέπει να εργαστούν με μεγαλύτερη ένταση. Και κυρίως Κάτι το οποίο φάνηκε είναι πως οι γνώσεις μας είναι υπερβολικά γενικές. Το 2050 είναι ένας χρονικός ορίζοντας που δεν απέχει τόσο πολύ για όλους μας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή, παρόλο που εγώ τότε θα είμαι 92 χρονών, οπότε μάλλον δεν θα προλάβω τη συζήτηση. Ελπίζω βέβαια ότι εσείς οι υπόλοιποι θα έχετε καλή υγεία και την δυνατότητα και τότε κάτι να κάνετε. Θα ήθελα όμως να δώσουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, ε, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν, μπορούμε με τον τρόπο αυτό να πλαισιώσουμε και τα λεγόμενά σας. Και θα μπορούν τα παραδείγματα αυτά να ε, χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς στο διάλογο που γίνεται. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τα απόβλητα είδη ηλεκτρονικών, ε, ηλεκτρονικών ειδών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Πόσα άτομα ε, ασχολούνται με το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ποια είναι η θέση τους. για να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια βιομηχανία που εργάζεται, ε, που με όταν έχουμε μια βιομηχανία εξορρυκτική ε, στην ε, Σουηδία, χρησιμοποιεί κάποιες από, κάποιον από τον εξοπλισμό της για να τον κάνει ανταλλακτικά για κινητά τηλέφωνα. Είναι ένα είδος ανακύκλωσης αυτών των ηλεκτρικών συσκευών. Ξέρετε πως στην Ουγγαρία, στο Μπουρούς πρόσφατα έγινε μια ε, φυσική καταστροφή μεγάλη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε το το ρηκτό το οποίο διαχύθηκε όμως τότε στην περιοχή που ήταν ευοξήτης δεν αποτελεί μόνο ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά μπορεί να αποτελέσει ε, και ένα ε, ορυκτό το οποίο μπορούμε να ανακυκλώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες ανακύκλωσης έτσι ώστε να γίνεται και βιομηχανική εκμετάλλευση όλων αυτών των ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Νομίζω ότι εξετάζοντας αυτές τις διαστάσεις θα δώσουμε κάποια θετικά παραδείγματα που θα πλησιώσουν τις προσπάθειες που κάνετε και έτσι δεν θα συμμετέχουν μόνο οι ηγέτες στην ε, λήψη αποφάσεων, αλλά θα δείξουμε και στους πολίτες πως είμαστε φιλόδοξοι στο θέμα αυτό της ε, ανακύκλωσης όλων αυτών των ειδών και εξοπλισμού, έτσι ώστε να κατακτήσουμε τους στόχους που αναφέρατε στην ε, παρουσία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Για την ε, ατζέντα του 2020 ε, και για τους πέντε στόχους εκεί, ε, πιστεύετε ότι πρόκειται να τους πετύχουμε και σας, ρωτώ το, και σας ρώτησα, γιατί αν δούμε ποια είναι, ποιοι είναι οι στόχοι κάθε κράτους μέλους για το 2020, θα διαπιστώσουμε ε, πως πολλοί έχουμε μείνει τόσο πίσω που δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους γενικότερους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αποδοτικότητα λοιπόν, ρωτώ, τα κράτη-μέλη έχουν ήδη όλα οριοθετήσει στόχους. Τους έχουν ποσοτικοποιήσει. Γιατί αν όχι θα ήθελα να μου πείτε ποιοι δεν το έχουν κάνει και πώς θα καταφέρουμε οι στόχοι αυτοί ε, να γίνουν δεσμευτικοί. Όσο για τα απόβλητα αυτά, είμαι εισηγητής για τα βιοαπόβλητα και η έκθεση αυτή το 2010 τον Ιούνιο εγκρίθηκε. Ρωτώ λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο να προχωρήσει στο θέμα των βιοαποβλήτων γιατί αποτελούν το 30% των αποβλήτων ε, που θάβονται. Θα κάνετε κάποιο είδος διαχωρισμό, κομποστοποίηση, έχετε προτάσεις που θα προστατέψουν τα εδάφη μας με τον τρόπο αυτό. γιατί είναι τεράστια τα ποσά που χρειάζονται για την ανακύκλωση κάθε χρόνο και με τον τρόπο αυτό αν κάναμε περισσότερες προσπάθειες πιστεύω ότι θα προχωρούσαμε προς μια κοινωνία με καλύτερες επιδόσεις ε, στην ανακύκλωση, κάτι που θα βοηθούσε στο να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Και ρωτώ το εξής, πώς είναι δυνατόν σε μια οδηγία ε, να μην έχουμε βάλει κανόνες για αυτή την κομποστοποίηση υψηλής ποιότητας τουλάχιστον ε, κανόνες που να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε τα κράτη-μέλη όχι μόνο να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε προηγούμενες οδηγίες αλλά πραγματικά η κομποστοποίηση να είναι υψηλής ποιότητας. Και να κάνω μια ακόμα ερώτηση η οποία συνδυάζεται με τις προηγούμενες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πώς θα ε, καταφέρει οι προτάσεις αυτές ή μάλλον η νομοθεσία η οποία θα απορρέει από αυτές και οι στόχοι να είναι δεσμευτικοί. Πολύ ωραία. Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος των ομιλητών. Έχουν ζητήσει ακόμα δύο τον λόγο, ο Κάρλος Σλούτα και η Άνια. Εφόσον μιλάμε για την ε, επάρκεια των φυσικών πόρων, Στη Σουηδία, στα μέσα του 19ου αιώνα, ανακαλύψαμε σπάνιες γέες. Τώρα, θα ενταθεί περαιτέρω η διαμάχη για αυτό το υλικό. Ε, πρέπει να γίνουν ανασκαφές σε βάθος για να αποκτήσει κανείς ε, ικανοποιητικές ποσότητες. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία και στην πολιτική ασφάλειας. Δηλαδή, αν δεν το πράξουμε αυτό θα προκαλέσουμε συγκρούσεις ανά τον κόσμο και αυτό είναι κάτι που υπόψη. Υπάρχουν όμως και όρια. Ας πούμε, τι είδου μέτρα προτίθεστε να λάβετε τι είδου φορολογία θα επιβληθεί ή αν θέλετε τέλος εξόριξης. Ε, και αυτό θα ήταν καλό, γιατί όχι, να πληρώνουν κάποιες εξορικτικές εταιρείες. Επίσης, κατά την άποψή σας, πού είναι τα όρια. Το αυτοκίνητο του 1914 του παρελθόντος χρησιμοποιούσε περισσότερη ενέργεια από σήμερα, αλλά όχι και πολύ μεγάλη διαφορά. Ο πρώτος μου υπολογιστή του 82 χρησιμοποιούσε 40 βατ και σήμερα ο δικός μου χρησιμοποιεί 80 βατ. Το διπλάσιο βεβαίως και είναι πολύ πιο γρήγορος, αλλά Εάν ε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να αποκτούμε όλο και περισσότερα, κάπου θα υπάρξει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να αποφασίσουμε για μια οικονομία η οποία δεν θα αναπτύσσεται μόνο με την ε, χρησιμοποίηση των υλικών, κάπως αλλιώς. Γιατί εάν ισχύει αυτό σήμερα, καταλαβαίνετε ότι στο μέλλον θα χρειαστούν ακόμα περισσότεροι φυσικοί πόροι. Και το μετά από 500 χρόνια θα είναι ασύλληπτο το ποσό, η ποσότητα που θα χρειαζόμαστε και πώς θα τον πετύχουμε αυτό το στόχο. Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα πώς μπορούμε να αποφασίσουμε για τη χρήση ενός οικονομικού συστήματος που δεν θα προκαλεί την ανεργία, οποτεδήποτε δεν υπάρχει ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την καινοτομία και να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο οι φυσικοί πόροι που υπάρχουν, τότε τι θα πούμε στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημα σε οικονομικό επίπεδο που υπάρχει και θα ήθελα να γνωρίζω την απάντησή σας επ' αυτού. Αυτό είναι πραγματικά το ερώτημα υπερπάντων και από εκεί απορρέουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και διάφορα εργαλεία που έχουμε. Κύριε Επίτροπε, έχω να σας υποβάλω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ακούσαμε ότι το 2013 θέλετε να το ανακηρύξετε σε έτος ε, ποιότητας της ατμόσφαιρας. Εγώ ε, είχα πριν από λίγο καιρό ηγήθηκα των ε, διαπραγματεύσεων από την πολιτική ομάδα για τις ρηπογόνε ρηπογόνες για τα ρούμενα σωματίδια και για τα συναφή. Και τότε είχαμε πει ότι τις εκπομπές ε, πρέπει να τις καταπνίξουμε στην πηγή, εν τη γενέση. Ε, και να θεσπιστεί και η σχετική νομοθεσία. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς, οι πόλεις, ε, οι μεγάλες πόλεις στα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν καμία δυνατότητα να τηρούν τις οριακές τιμές, κυρίως όσον αφορά τις τιμές NOx περί αζότου. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι προτείνεται να κάνει η Κομισιόν στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Δηλαδή, ίσως ε, η πλειοψηφία των ε, κρατών μελών να μην τηρήσει αυτές τις ε, νέες ανώτατες τιμές. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε τι προτείνεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, από ό,τι βλέπετε υποβλήθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις και σας εκφράστηκε και υποστήριξη από την Επιτροπή μας. Κανείς βέβαια στην Επιτροπή δεν μπορεί να είναι αντίθετο με επαρκείς φυσικούς πόρους στην Ευρώπη. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό και πώς θα εφαρμοστεί περαιτέρω ο χάρτης πορείας. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αλλά από ό,τι βλέπω σημειώσατε αρκετά πράγματα. Θα περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. Ίσως λοιπόν πρέπει να ξεκινήσω με μια γενική απογραφή της κατάστασης και να δούμε ποιες μπορεί να είναι και οι εξελίξεις μελλοντικά και κατόπιν θα απαντήσω και σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αν παρακολουθήσουμε το τι συνέβη στον 20ο αιώνα και ποιες είναι οι προθέσεις μας για τον 21ο, και κυρίως αν λάβετε υπόψη πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ε, βασιζόμαστε στις εισαγωγές για όλους αυτούς τους πόρους, όπως επίσης αν δείτε την εξέλιξη σε επίπεδο τιμών, τότε ναι, Σίγουρα κυριάρχησε ε, στον 20ο αιώνα, ε, κυριάρχησαν οι πόροι, ε, οι φθηνοί πόροι. Για τον 21ο αιώνα η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Οι τιμές λοιπόν αυτών των ειδών έχουν αυξηθεί και οι περισσότερες επιχειρήσεις για τα επόμενα πέντε έτη θεωρούν πως οι τιμές αυτές θα αυξηθούν παραπάνω. Όταν λοιπόν Μιλάμε για παγκόσμιες εξελίξεις, για εξάρτηση από τις εισαγωγές, για διακύμανση των τιμών προς τα επάνω, τότε διαπιστώνουμε πως η διάθρωση του κόστους για τις περισσότερες επιχειρήσεις επιβαρύνεται πολύ περισσότερο από την απόκτηση των πρώτων υλών από ότι από το εργασιακό, από εργασιακό κόστος. Άρα λοιπόν το να είμαστε αποδοτικοί στη χρήση των πόρων που έχουμε ε, δεν ε, θα εξασφαλίσει μόνο ένα καλύτερο περιβάλλον μελλοντικά, αλλά θα βελτιώσει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και οι μεσαίες επιχειρήσεις το έχουν κατανοήσει αυτό. Νομίζω το μήνυμα έφτασε πριν από τον αγγελιοφόρο και το κάνουν γιατί από αυτό εξαρτάται η ίδια τους η επιβίωση. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήσεις που έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη άποψη για το τι συμβαίνει και βασίζουν τη στρατηγική τους σε κάποιες ουσιαστικές μεγάλες τάσεις, μία από τις οποίες διαφαίνεται σήμερα και η οποία είναι το να είσαι κανείς πιο αποδοτικός. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση γύρω μας. Το βασικό πρόβλημα είναι το πώς θα μπορούσαμε εμείς να εντάξουμε στη δική μας διαδικασία χάραξης πολιτικής το θέμα αυτό έτσι ώστε να είμαστε εμείς στην εμπροστοφυλακή και να παρακολουθήσουμε και να συνοδεύσουμε τις επιθυμίες του βιομηχανικού κλάδου. Γιατί πολλές από τις ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τη βιομηχανία έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή γιατί βεβαίως έχουν ε, ως στόχο την προστασία του status quo. Αυτό βεβαίως δεν θα τους εξασφαλίσει ανταγωνιστικότητα στο μέλλον, αλλά υπάρχουν ε, και κάποιες κοντόφθαλμες πολιτικές, τις οποίες εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω πως ε, αν σταθούμε ένας δίπλα στον άλλο και πιέσουμε όλοι μαζί έτσι ώστε αυτό να γίνει το κοινό μας σύνθημα θα τα καταφέρουμε. Διαφορετικά θα μείνουμε πίσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο τελικός μου στόχος. Δηλαδή, σε όλους τους κλάδους στους οποίους αναφερθήκατε, σε όλους κάτι συμβαίνει. Κάποιες εξελίξεις τρέχουν. Όμως, χρειαζόμαστε ένα κίνημα το οποίο θα στηρίξουμε ε, επίμονα ε, υπομονετικά, με νομοθεσία, με πρότυπα, με μετρήσεις, με στοιχεία, για να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε όλοι. Άκουσα και την ερώτηση της φίλης Λουίζα... Νομίζω πως ακολουθούμε τη σωστή διαδρομή. Όμως, και θα είμαι ειλικρινής εδώ. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητάμε πιο πολύ τα προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης από ότι συζητάνε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων το θέμα του περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φανούμε θαραλέοι και όταν συζητήσαμε το θέμα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος πρόσφατα είπα στους συναδέλφους ότι στο ΕΚΟΦΗΝ δεν συζητάνε τα δικά μας προβλήματα του περιβάλλοντος, ενώ εμείς όταν συζητάμε θέματα περιβάλλοντος πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη τη διάσταση ε, θέσεων εργασίας και ε, ανάπτυξης. Αν λοιπόν το προσπαθήσουμε όλοι μαζί, κάτι θα καταφέρουμε. Ε, ε, ζούμε μια εποχή κρίσης και δυστυχώς για να είμαστε ρεαλιστές είναι πολύ πιο δύσκολο να συζητήσουμε και να προωθήσουμε το θέμα μας και αυτό συγκρίνοντας με άλλες εποχές μεγαλύτερης αυθονίας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε ε, να μπούμε κι εμείς στη συζήτηση των οικονομικών θεμάτων πείθοντας πως μπορουμε να μπουμε και εμεις στη συζητηση των οικονομικων θεματων πειθοντας πως ειναι και οικονομικά τα ωφέλη ε, με το να γίνουμε πιο αποδοτικοί και έτσι θα εξασφαλίσουμε και περιβαλλοντολική προστασία για το μέλλον, αλλά και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε όμω όλοι να συμφωνήσουμε τι λεπτομέρειε, το καταλαβαίνω. Θα πρέπει όμω να συμφωνήσουμε τουλάχιστον μια πολιτική συνεκτική και μια γενικότερη κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Και θα ήθελα εδώ να διατρέξω μία-μία τι ερωτήσει. Για τη θετική χρειά που μπορούμε να δίνουμε, ναι, νομίζω ότι Καλό είναι να δείχνουμε αισιοδοξία. Τώρα, την οδηγία, τον κανονισμό, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και εγώ ο ίδιος. Γιατί καμιά φορά δεν μεταφέρουν ε, τις οδηγίες στα κράτη-μέλη με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Μία βασική απάντηση που μπορώ να δώσω είναι ότι εμείς μεν συμφωνούμε τις κατευθύνσεις, αλλά τα κράτη-μέλη βεβαίως γνωρίζουν καλύτερα ποια είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία που μπορούν να ανταποκριθούν στις δικές τους συγκεκριμένες περιστάσεις. Η ερώτηση όμως που υποβάλλατε νομίζω ε, γίνεται όλο και πιο σχετική. Μιλήσατε για επιδοτήσεις. Ίσως εδώ πρέπει να πω δύο λόγια. Μιλάμε για το εξάμεινο και μάλιστα σήμερα ε, δημοσιεύθηκε αυτή η ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη και βέβαια κάνω ό,τι μπορώ, αλλά το περιβάλλον και τα επιχειρήματα για την αποδοτικότητα δεν μπορούν να τονιστούν παραπάνω από ότι ήδη υπογραμμίζονται. Εγώ προσπαθώ να πιέσω προς τρεις κατευθύνσεις. Καταρχήν, φορολογία. Όταν λέμε φορολόγηση, μιλάμε για ε, συστάσεις που θα απευθύνουμε ε, στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, να μην φορολογείται τόσο πολύ η εργασία όσο η πόρη. Αυτό είναι μια σύσταση και να το λάβουν υπόψη στο εθνικό φορολογικό σχέδιο. Μόνο τόσο μπορούμε να πούμε. Δεν είμαστε αρμόδιοι για φορολογική πολιτική, αλλά βεβαίως αποτελεί τμήμα των κοινών προσπαθειών. Και αυτό συμβαίνει και για τις επιδοτήσεις που είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. Δεν ξέρω αν ε, εσείς το γνωρίζετε, αλλά για τα 45 δις ε, που δαπανούν οι επιχειρήσεις. Για τον εταιρικό στόλο καταλαβαίνετε ότι εκεί θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ τις επιδόσεις μας. Και έχω και πολλά τέτοια παραδείγματα ακόμα να δώσω. Θα ήθελα να δούμε βέβαια και το θέμα της ενέργειας έτσι ώστε να ακολουθήσουμε μια πιο συγκροτημένη προσέγγιση, η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σταδιακά. Και για το τρίτο θέμα στο οποίο πιστεύω πως θα πρέπει να σταθούμε, είναι η εσωτερική αγορά για τα περιβαλλοντικά αγαθά, όπου θα έχουμε βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Νομίζω ότι και αυτό θα έπρεπε να μπει ε, στο διάλογο. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα ακολουθήσουμε τα όσα σας περιέγραψα. Ποιο είναι το όνειρό μου. Όταν προτείνουμε, ε, όταν μάλλον παρουσιάσει ο κύριος Ρεν την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη και επίσης όταν ο Επίτροπος Άντορ ε, αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί, να είμαι κι εγώ εκεί. Για να μιλήσω για το περιβάλλον. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει κάτι τέτοιο, αλλά ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Τώρα, Λίντα, για το κατά πόσο οι άλλες επιτροπές κάνουν κάτι αντίστοιχο και αν διαβολευόμαστε για τα θέματα αυτά, εγώ προσπαθώ με οργανωμένο τρόπο να συνεργάζομαι με όλους αλλά πολλές φορές με κατηγορούν ότι πλατιάζω, γιατί βέβαια δεν είναι εύκολο να είσαι στοχευμένος όταν μιλάς για πολλά θέματα. Για την κοινή γεωργική πολιτική, για την αλληλεία, για τη συνοχή. Και μπορώ να τα πω και μαζί σας αν το επιθυμείτε, αλλά νομίζω ότι εκεί τα έχουμε πάει πολύ καλά έχουμε καταφέρει το θέμα του περιβάλλοντος να το εντάξουμε σε όλες αυτές τις πολιτικές. Και στην βιοπικιλότητα και στα υπόλοιπα πλαίσια ε, για το καθαρό νερό κτλ. Πιστεύω ότι ήμασταν αποτελεσματικοί. Βέβαια, θα ήθελα να περάσω και από την Επιτροπή Ήτρε, όπως επίσης και από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού αλλά δυστυχώς στο Συμβούλιο αυτό δεν κατάφερα να πάω γιατί συνέβη κάτι πολύ παράξενο το οποίο δεν θα σας διηγηθώ. Εν πάση περιπτώσει πήγα και στην ε, Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου και πρέπει να σας πω πως δεν θα είμαστε ποτέ ε, επιτυχημένοι στην προσπάθειά μας εάν δεν ε, κάνουμε μια οριζόντια προσπάθεια γιατί αν συζητάμε τα θέματα αυτά μόνο μεταξύ μας μικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιοριζόμαστε στα θέματα του χαρτοφυλακίου μας, του Συμβουλίου μας, της Επιτροπής μας, αλλά θα πρέπει να βγούμε εκτός, γιατί για το περιβάλλον, αν θέλω να το βελτιώσω, θα πρέπει να αντιμετωπίσω το θέμα της ενέργειας, των μεταφορών, οποιαδήποτε άλλη πολιτική ή βιομηχανικός κλάδος εμπλέκονται. Αν λοιπόν δεν δράσουμε εκεί, δεν θα τα καταφέρουμε. Για το σχιστολιθικό αέριο μιλήσαμε για τους κινδύνους ε, ε, που μπορεί να δημιουργήσει, ε, που μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση σε καύσιμα στην Ευρώπη και μιλήσαμε και για κάποιες μελέτες οι οποίες γίνονται για να δούμε ποια θα είναι η υπερβαλλοντολική επίπτωση της χρήσης αυτού του αερίου αλλά και της εξόρυξης αυτού του αερίου. Και θα δούμε για κάποιες χημικές ενώσεις επίσης που χρησιμοποιούνται στην υδραυλική εξόρυξη εάν ε, προκαλούν πρόβλημα και θα δούμε και για το σχέδιο για αυτό το νέο αέριο μπορούμε ε, να εντάξουμε ό,τι έχουμε εντάξει στα υπόλοιπα για τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες. Για να δούμε και για το REACH το θέμα που θίξατε είναι κατά πόσο θα έπρεπε και κάποιες ακόμα ουσίες να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για αδειοδότηση. Όλα αυτά βρίσκονται στα σκαριά. Μαζεύουμε πληροφορίες, συλλέγουμε στοιχεία και θα σας εξασφαλίσω πως οι εξελίξεις εδώ θα εξεταστούν με ιδιαίτερη σοβαρότητα και από μένα αλλά και από τις υπηρεσίες μου. Ε, αδειοδότηση για την ουσία την οποία αναφέρατε. Η αρχική μου αντίδραση είναι πως θα έπρεπε όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο κατάλογος αυτός να είναι πλήρης. Το είπα και με τον Επίτροπο κύριο Τατζάνη. 136 ουσίες μέχρι το τέλη της επόμενης χρονιάς. Και έχω και την συνάντηση αύριο νομίζω το μεσημέρι για το μήνυμα που θα στείλω στη ΣΑΦΕΚ γιατί θα πρέπει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε να είναι ελεγχόμενο. Και όσο, το όσο πιο γρήγορα γίνει η υποκατάσταση, η αντικατάσταση αυτών των ουσιών που θα έχουμε στον κατάλογο, τόσο καλύτερα. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Επιστημονική Επιτροπή να εξετάζει μόνο ε, ποιε, αλλά και το πότε θα γίνει αυτή η υποκατάσταση. Και επαναλαμβάνω, εάν υπάρχουν βλαβερές ουσίες, η αντικατάσταση αυτών θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα από τα θέματα που έχουμε στον οδικό χάρτη για την αποδοτικότητα στην ενέργεια είναι όλες αυτές μέχρι το 2020 να έχουν τοποθετηθεί στον κατάλογο και να έχουν υποκατασταθεί. Τώρα για την επιχειρηματική πολιτική νομίζω και στην παρουσίαση που σας έκανε εισαγωγικά σας μίλησα για διάφορα θέματα και οι φήμες για αναβολή του οδικού χάρτη κατά τη γνώμη μου είναι απλώς φήμες, δεν έχω ακούσει κάτι αντίστοιχο. Η κυρία Ρόσμπαχ μου ρώτησε κάτι για τα τρόφιμα τα οποία πετάμε και δεν ξέρω Αν είδατε μια δράση που ξεκινήσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, πήγα σε δύο-τρεις χώρες για τα εγγένεια αυτής της δράσης, η οποία είναι πολύ, ε, πολύ αποτελεσματική, εστιάζει στη νέα γενιά και στις νέες οικογένειες, που έχουμε αυτές τις σακούλες σούπερ ε, οι οποίες ε, βγάζουν αυτό το, το τραγουδάκι που λέει ότι πρόσεχε τι αγοράζεις, πρόσεχε γιατί πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένο καταναλωτής είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην προσπάθεια να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Για το ευρωπαϊκό εξάμεινο Έχουμε την ε, οδηγία για την ενεργειακή, φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων, όπου όμως τα πράγματα πάνε αργά. Θα χρειαστούμε χρόνο. Εάν περάσουμε μέσω της οδού των εθνικών συστάσεων, τότε θα πρέπει τα εθνικά προγράμματα να εντάξουν κάποια τέτοια μέτρα, το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό. Βιομάζα. Ακόμα και αν δεν συνδέεται άμεσα με το χαρτοφυλάκιο μου, παρακολουθούμε συνέχεια το θέμα, έτσι ώστε τα κριτήρια ε, βιωσιμότητας να συμπεριλαμβάνει το θέμα αυτό. Βέβαια έχουμε τους επιτρόπους Ότιγκερ και Χίλντεργαρτ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης και όπως είπατε και εσείς χρειαζόμαστε αυτά τα κριτήρια βιωσιμότητας τα οποία είναι το α και το ω. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η λογική η οποία θα κυριαρχήσει. Ο Καρλ Γιατί επιλέξαμε αυτή την προσέγγιση, γιατί πέρυσι δεν μπορούσαμε να δώσουμε τις δύο μάχες ταυτόχρονα. Επιλέξαμε λοιπόν ένα ευρύτερο πεδίο μάχης. Το οποίο βέβαια μας κόστησε με κάποια από τα εφαρμοστικά μέτρα μετά. Διαφορετικά συμφωνώ με τις όσες παρατηρήσεις κάνατε. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και βέβαια θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή για τα ύδατα κοιτάμε ε, τις βασικές παραμέτρους. Του χρόνου θα είναι ένα από τα θέματα που θα μας αποσχολήσει. Έχουμε επίσης και το Eco Design και αυτό θα σχολιάσω αργότερα. Τώρα για την εφαρμογή, όντως θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε τις ε, προσπάθειές μας. Ελπίζω λοιπόν ότι στην εφαρμογή του εβδόμου πλησίου θα κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Judith, ε, όσον αφορά τους ε, στόχους ανακύκλωσης κατά πόσο θα υπάρχει ενημέρωση ή όχι κατά και το εξαμήνου. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα σύστημα ενημέρωσης σε, τακτά χρονικά διαστήματα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα επ' αυτού. Ε, το πρόβλημα είναι περισσότερο ότι δεν καλύπτονται κάποιοι από τους στόχους ε, που ανέφερα. Εμείς λοιπόν προτιθέμεθα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε ε, κάποιες, ε, κάποιοι στόχοι στο τομέα των αποβλήτων πράγματι να επιτευχθούν. Ε, σε γενικές γραμμές όμως, όπως σας είπα, ακολουθούμε τη στάση των στόχων και των δικτών. Και έτσι το 2013 πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα. Τώρα, σαν αφορά την απαγόρευση χώρων ανοιχτής ταφής. Αυτή τη στιγμή αγωνίζομαι με το πώς θα μπορέσουμε να απογορεύσουμε παράνομους τέτοιους ε, χώρους. Ορισμένα προβλήματα εξακολουθούν να έχουν Ορισμένε χώρε με εξακολουθούν να έχουν ε, σοβαρά, σοβαρά προβλήματα διαχείριση αποβλήτων. Έχουμε πέντε χώρε που πλησιάζουν αυτό που θα επιθυμούσατε, αλλά και σε αυτέ τι χώρε το πρόβλημα είναι ε, τι γίνεται με την καύση. Η καύση δεν θα πρέπει να είναι η ε, πρακτική αμέσως μετά τις ε, χωματερές. Εμείς επιθυμούμε ε, να προάγουμε την ανακύκλωση και να μειωθούν γενικά, μειωθεί γενικά ο όγκος των αποβλήτων. Τώρα, όσον αφορά την απαγόρευση εξαγωγής αποβλήτων, ε, πράγματι, ε, προσέχουμε, έχουμε στέψει την προσοχή μας στις δευτερογενείς αγορές της Ευρώπης ε, σε ορισμένους τομείς παρήματος χάρη στο Χάλιβα εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες διαμαρτυρίες για εξαγωγές είμαι όμως σίγουρος ότι μπορούμε να κρατήσουμε την κατάσταση υπό έλεγχο και έτσι λοιπόν ε, θα εξετάσουμε και το πρόβλημα που αναφέρατε. Όσον αφορά στην ιεράρχηση των πρώτων λόγων, ακόμα δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο αυτό που είπε ο Καρλ Χάιντς. Δηλαδή να εφαρμόσουμε εκείνα επί των οποίων ελπίζουμε να συμφωνήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι η επάρκεια πόρων είναι πρόταση της Κομισιόν. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε και τη στήριξη των κρατών μελών ε, και είμαι σίγουρος ε, βέβαια ότι εσείς θα κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και εκεί θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Κρήτονα. Αν θεωρούσα ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι, θα παρακολουθούσα το κατά πόσον πλησιάζουμε το στόχο ή όχι το θέμα δεν είναι να πούμε τώρα είμαστε σε καλύτερη θέση από ότι πριν από λίγο καιρό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ορισμένα μέτρα που ελήφθησαν στην κοινή γεωργική πολιτική και την κοινή πολιτική αλίες αναμφίβολα ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αναρκεί αυτό, αυτό είναι δύσκολο να το πούμε. Ίσως ε, πράγματι ε, πρέπει να γίνουν και άλλα πολλά, αυτό είναι πιο τίμιο να το πούμε. Και κάτι που ε, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας η νομοθεσία για τα ξένα είδη. Όμως εδώ πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία. Είναι δύσκολο να πούμε ένα χρόνο ε, μετά την Αγκόγια κατά πόσο να έχουμε προχωρήσει όχι. Έχουμε την ε, σωστή στρατηγική, έχουμε τους, ε, τη στρατηγική και τους στόχους το Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή συζητάμε για τη δράση με το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα γενικά είναι πολύ καλή. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό που αφορά στην ένταξη, συμπερίληψη στην κοινή γεωρική πολιτική και την πολιτική αλίας. Τι πρέπει να γίνει πρώτα ε, και κατά πόσον το περιβαλλοντικό ε, συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο να προχωρήσει στον τομέα του πολιτούς ε, πλαισίου χρηματοδότησης. Πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι το, ο στόχος αυτών που υποσχεθήκαμε στην Αγκόγια. Στον κύριο Άντερ απευθύνομαι. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία που είπατε, που αναφέρατε, αυτήν θα την προσυπέγραφα χωρίς ε, κανένα πρόβλημα. Η ανακύκλωση είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς με την ανακύκλωση μπορεί κανείς ε, να καταλήξει σε εναλλακτικέ λύσεις που είναι πολύ καλύτερες από το να αρχίζει κανείς την ε, εξόριξη και μάλιστα υπό συνθήκες που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου ασφαλείς. ή αν δεν το πούμε έτσι, να το πούμε αλλιώ, να πούμε ότι δεν είναι και τόσο αυτόες οι συνθήκες αυτές. Πράγματι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της επεξεργασίας τοξικών ουσιών. Κύριε Φερνάντες, αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας. Αυτό δεν εμπίπτει άμεσα στις δικές μου τις αρμοδιότητες, όμως πρόσφατα εγκρίναμε ένα έγγραφο το οποίο ε, έχει ως στόχο να κλείσει το κενό που υπάρχει. Και από τη συζήτηση που έλαβε χώρα θυμάμαι αναφέρθηκε ότι η Κομισιόν θα εξετάσει το κατά πόσον μπορεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της δέσμευσης. Βιοαπόβλητα απόβλητα τώρα. Ε, νομίζω έχω επανειλημμένα αναφερθεί στους στόχους και έχω εξηγήσει και τους λόγους ε, γιατί δεν χρειαζόμαστε μία ειδική οδηγία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ε, δεν ε, σκοπεύουμε να εκδώσουμε οδηγία για τα βιοκαύσιμα. Το σκεφτόμαστε. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Ορισμένα κράτη-μέλη ήδη σήμερα τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Έχουν ήδη νομοθεσία που δεν είναι δεσμευτική, αλλά κανείς δεν τους εμποδίζει να την μετατρέψουν δεσμευτική και τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Αυτή η στόχη λοιπόν είναι υπό ως προς την καινοτομία, κοιτάξτε, έχουμε όταν ε, ασχολούμεθα με την παραγωγή και με την κατανάλωση, στην ε, παραγωγή ε, αναμφίβολα οικολογικό σχεδιασμός. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Γνωρίζω ότι μερικοί φοβούνται ότι αυτό, δηλαδή προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα στην ενέργεια θα φτάσουμε σε ένα γραφειοκρατικό τέρας, αλλά τελικά αν κατά τη διάρκεια, στη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος σκεφτεί κανείς τι υλικό θα χρησιμοποιηθεί, πώς θα παραχθεί και πώς θα γίνει ανακύκλωση, νομίζω το πρόβλημα λύνεται. Μετά, ε, όσον αφορά την, ε, τις οικολογικές ετικέτες και την ενημέρωση του καταναλωτή, εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, εκατοντάδες ετικέτες που δεν θα τις καταλαβαίνει κανείς, να είναι ευανάγνωστες και να βοηθούν τον καταναλωτή να αποφασίσει σωστά. Καινοτομία, η καινοτομία έχει αποδείξει επανολωμένα ότι ε, μπορεί να πετύχει ε, πολλά περισσότερα από αυτά που εμείς προσδοκούμε. Ο ε, Μάλθους ε, είπε πριν από χρόνια ότι υπάρχει ο πληθυσμός γης είναι πεπερασμένος και υπάρχει και η εξή ιστορία. Τότε όταν είχαν παλιά τις άμαξες ήθελαν να τις καταργήσουν γιατί οι κοπριές ε, δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα. Αυτό ήταν ένας λόγος. Και επίσης θυμάμαι ε, κάποια προφητεία σε εισαγωγικά που είχε πει ότι το 92 δεν θα υπάρχουν πλέον καύσιμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να ε, πιέσουμε την ε, πολιτική που ακολουθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό το συζητάει η Κομισιόν. Ούτε προσπαθώ να πω ότι δεν θα πρέπει να εξετάσουμε την ε, αντίδραση. Γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε από κοινού και την προσφορά και τη ζήτηση. Απλά θέλω να πω ότι ενδέχεται να εκπλαγούμε όσον αφορά την καινοτομία. Και αν δώσουμε τα σωστά μηνύματα, ε, οπωσδήποτε θα πάρουμε και τις σωστές απαντήσεις μέσα από την καινοτομία. Πιστεύω λοιπόν ότι η βιομηχανία χρειάζεται ένα σαφές μήνυμα και αυτό το αποκτά ε, από το δικό της το χώρο, ότι θα πρέπει να μετακινηθεί στη σκέψη, δηλαδή από την παραγωγικότητα εργασίας στην παραγωγικότητα των πρώτων υλών. Αυτό είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Και τέλος όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Πράγματι, έχουμε πρόβλημα με την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν πολλά θέματα που εκκρεμούν και εγώ ε, ξεκίνησα τη συζήτηση με το Κολέγιο των Επιτρόπων στις αρχές του έτους ε, γιατί χρειάστηκα την υποστήριξή τους. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το λύσω χωρίς την ε, υποστήριξη ε, του Επιτρόπου Μεταφορών, ε, Αλίας και άλλων, όλων των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Καταλήξαμε λοιπόν σε μια συμφωνία, δουλεύουμε πάνω σε αυτές τις προτάσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα του ε, των οξυδίων αζότου ας πούμε έχουν ε, εξαφανιστεί κάθε άλλο. Είναι σοβαρά προβλήματα στον τομέα των μεταφορών. Εστιάζουμε την προσοχή μας στις ε, μετρήσεις και μετά στις εκπομπές ε, εκεί πιέζουμε λιγάκι τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει κατά κύριο λόγο να διατρέχει τις ε, σκέψεις μας είναι η υγεία των πολιτών. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Ο ΠΟΗ μας ε, στέλνει το μήνυμα ότι τα οι προδιαγραφές που έχουμε σήμερα ίσως θα πρέπει στο μέλλον να καταστούν περισσότερο αυστηρές αν δούμε τη γνώση που έχουμε συγκεντρώσει εδώ και χρόνια η οποία δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση ανάμεσα ε, στην υγεία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας θέλω να ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και επίσης ε, πολύ σοβαροί είμαστε, κάνουμε δουλειά μας και όσον αφορά τις ε, παραβάσεις. Γιάννη Ποτόσνη, κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι η δέσμευσή σα ε, είναι σίγουρη ε, και είχατε το χρόνο να μας δώσετε προσωπικές απαντήσεις ε, σε όλα τα ερωτήματα των βουλευτών και να μας παρουσιάσετε το όραμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την αφοσίωσή σας και για τη δέσμευσή σας. Βλέπετε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχετε σαφή υποστήριξη θα πάτε στις άλλες επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου και θα τους πείτε ότι μιλήσαμε πολύ για την ανταγωνιστικότητα και για τις ε, βιομηχανικές δυνατότητες, ε, ούτως ώστε να ενδιαφερθούν και εκείνοι για την διατήρηση του οικοσυστήματος και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη αυτή η συζήτηση και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει για την έκθεση που θα εξετάσουμε. Θα παρακολουθούμε τις συζητήσεις ε, που θα συνεχίσετε εσείς ε, για το θέμα της ένταξης ε, του θέματος της αποτελεσματικότητας των πόρων σε όλες τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε και στο επανειδήν. Okay, then we straight away... Λοιπόν, περνάμε κατευθείαν στην έκθεση Γκέρμπεν Γιάν και Μπράντι για το ίδιο θέμα. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους φόρους. Αφού τώρα έχουμε κάνει τόσο μακρά συζήτηση για το ίδιο θέμα, νομίζω ότι μπορούμε να συντομεύσουμε ίσως τη συζήτηση που θα ακολουθήσει για την έκθεση. Σας ακούσουμε τον κύριο Γιάννη τι έχει να μας πει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ 32 λεπτά. Θα είμαι πολύ πιο σύντομος. Παρ' όλα αυτά, δεδομένη τη σημασία και τη ευρύτητα του θέματο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό το έγγραφο εργασία. Και ξεκινώ με τις σημερινές εφημερίδες. Αν δείτε το σημερινό τύπο, την πρώτη σελίδα θα δείτε ότι υπάρχει η οικονομική κρίση, η κρίση του ευρώ κλπ. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην μας τυφλώσει η οικονομική κρίση και χάσουμε τις πιο θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Και τις προηγούμενες ε, δύο ώρες της συζήτησή μας ακούσαμε ότι σε λίγα χρόνια θα φτάσουμε τα 9 δισεκατομμύρια ως πληθυσμό του πλανήτη μας. Και ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι όλο και περισσότεροι ε, πολίτες αποκτούν εισοδήματα μέσης τάξεως ε, με αντίστοιχες δυνατότητες κατανάλωσης. Ανέφερε ο Επίτροπος ε, τη λέσχη της Ρώμης και ένα έγγραφο του 1972 με αποκαλυπτικές συνέπειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πλανήτης μας είναι μικρός και δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, αλλά λόγω των θεμελιωδών αλλαγών είναι ξεκαθαρό ότι θα αλλάξει και η οικονομία ριζικά. Σπανίζουν πλέον οι πόροι και για γεωγραφικούς ή για πολιτικούς λόγους, δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι λόγοι, σπανίζουν πάντως ε, οι πόροι και γίνονται και περισσότερο δαπανηροί. Η σπάνιση των πόρων είμαι βέβαιος ότι είναι ε, μία από τις ε, βασικές αιτίες για την επανάσταση στο θέμα της οικολογικής αντιμετώπισης των πόρων. Άλλες αιτίε είναι η προτίμηση των καταναλωτών, γιατί βλέπετε όλο και περισσότερο ότι οι καταναλωτές θέλουν να καταναλώνουν με τρόπο που να συντείνει στην βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό το συνειδητοποιούν σιγά σιγά και οι κατασκευαστές και παραγωγοί. Και όταν έκανα και την ερώτησή μου στον Επίτροπο προηγουμένως, αυτό είχα κατά η αποτελεσματικότητα των πόρων δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε κατά μέρος, διότι τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Όχι βέβαια, πρέπει πολύ δραστήρια να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποτελεσματικότητας των πόρων, ακριβώς διότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Και αν το Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μήνυμα αυτό πρέπει να είναι ότι χρειαζόμαστε ε, να το αντιμετωπίσουμε με πολύ πιο έντονο και ε, έντονα επίγοντα χαρακτήρα από ό,τι μέχρι τώρα. Δεδομένης της ε, οικονομικής σημασία που έχει λοιπόν η αποτελεσματικότητα των πόρων, για μένα είναι προφανές ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία για να αναζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το, πρόβλημα. Εμείς ως πολιτικοί δεν μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη χρήση των πόρων δρώντας χωριστά μακριά από τη βιομηχανία. Μαζί με τη βιομηχανία πρέπει να δράσουμε. Και γι' αυτό ζητώ από τη βιομηχανία να λάβει πιο συγκεκριμένη θέση από ό,τι μέχρι τώρα. Και έχω μιλήσει με πολλές εταιρείες, με πολλές ενώσεις και συνδέσμους βιομηχάνων τους τελευταίους μήνες και βλέπω ότι είναι δραστήριοι, αλλά δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολιτικοί και ως λαμβάνοντας αποφάσεις, ούτως ώστε να γίνει η Ευρώπη περισσότερο αποτελεσματική όσον αφορά την χρήση των πόρων. Και υπάρχουν εταιρείε οι οποίε ηγούνται ε, της πρωτοβουλία αυτή. Πολλέ εταιρείε κάνουν πολλά και επενδύουν πολλά στην αποτελεσματικότητα των πόρων, διότι το βλέπουν στην καθημερινή τους δραστηριότητα, πόσο σημαντική είναι η πόρη στην διάθρωση του κόστους και εστιάζουν σε αυτό. Υπάρχουν όμως άλλες εταιρείες που δεν έχουν πλήρη επίγνωση ή προσπαθούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και αυτή τη στάση τη βλέπουμε και στην Επιτροπή πολλές φορές το Κινέζικο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε, στην τελευταία του έκδοση ε, λέει ότι η Κίνα χρειάζεται περισσότερο ε, βιώσιμες επενδύσεις και αυτό θα οδηγήσει σε 9,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Κίνα. Το ίδιο πιστεύω ισχύει και για την Ευρώπη. Είναι ένα ισχυρό οικονομικό επιχείρημα και πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς σε αυτό τον τομέα και πρέπει να γίνουμε περισσότερο φιλόδοξοι και εμείς και οι εταιρείε. Χρειάζονται κίνητρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, τα κίνητρα θα πρέπει να μας οδηγούν σε καλύτερες υποδομές για τη χρήση των πόρων, ίσως δίνοντας και μεγαλύτερη νομική ευελιξία στις εταιρείε για να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια πολιτική αποτελεσματικότητα των πόρων, αλλά παράλληλα με τα κίνητρα χρειαζόμαστε και κυρώσεις. Αυτό θα μπορούσε να λάβει τη μορφή της φορολογίας ε, για να έχουμε και, το, τα κίνητρα αλλά και ε, ε, τις ποινές όπου χρειάζεται. Και πρέπει η Επιτροπή να εισαγάγει και συγκεκριμένους στόχους. Ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου να τονίσουμε τον επίγοντα χαρακτήρα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι στον τομέα των πόρων, διότι η δική μας ήπειρο είναι η πλέον εξαρτώμενη από τις εισαγωγές πρώτων υλών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Κάποια μεμονωμένα κράτη-μέλη προσπαθούν να εξασφαλίσουν την, τον εφοδιασμό τους, προσπαθούν να έχουν αποθέματα, αλλά η Ευρώπη συνολικά δεν βρίσκεται σε ηγετική θέση. Η Γερμανία καταβάλει πολλές προσπάθειες, παραδείγματος χάρη, προσπαθεί να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της σε σπάνιες γέες, αλλά γιατί να το κάνει μόνη της η Γερμανία αυτό. Γιατί να μην χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά που είναι ισχυρότερη και τι νόημα έχει να κάνει κανείς κάτι σε εθνικό επίπεδο, εφόσον η εμπορική πολιτική είναι ευρωπαϊκή πολιτική και όχι η πολιτική του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Σκέφτομαι διάφορα πολύ συγκεκριμένα μέτρα και ζητώ από τους συναδέλφους να τα εξετάσουν και να τα σχολιάσουν για να μπορέσω να τα συμπεριλάβω στο σχέδιο έκθεσής μου. Εξετάζουμε τα συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα της εμπορικής πολιτικής Υπάρχει η πολιτική των αποβλήτων και ορισμένα παραδείγματα ήδη αναφέρθηκαν στις ερωτήσεις που υπευλήθησαν στον Επίτροπο και στις απαντήσεις που έδωσε ο Επίτροπος. Και πιστεύω ότι η στρατηγική μας για τα απόβλητα εστιάζεται πάρα πολύ σε κάτι το οποίο πρέπει να ξεφορτωθούμε και όχι σε αυτό που πρέπει να δούμε, δηλαδή ότι τα απόβλητα έχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε θετικά. Οι Δήμοι και οι κοινότητες ε, δαπανούν πάρα πολλά χρήματα για την διάθεση των αποβλήτων, ενώ θα έπρεπε ε, να φροντίσουμε να βρούμε εταιρείε που θα πληρώνουν τους Δήμους και τις κοινότητες για να παίρνουν τα πολύτιμα υλικά ανακύκλωσης. Επίσης, ο οικολογικός σχεδιασμός είναι ένα σημαντικό τομέα. Θα πρέπει να θέσουμε στόχους για τον οικολογικό σχεδιασμό, γιατί αυτή τη στιγμή τα προϊόντα σχεδιάζονται με τρόπο τέτοιο που είναι αδύνατον να ε, αφαιρέσουμε τα πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά από αυτά τα προϊόντα. Άρα, ο οικολογικός σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός και είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας για το μέλλον. Για τους εταιρικούς στόλους δαπανώνται 54 δισεκατομμύρια ευρώ από ό,τι είδαμε στη σχετική έρευνα. Φανταστείτε να είχαμε περισσότερο ε, οικολογικά ε, σχεδιασμένα αυτοκίνητα, τι εξοικονόμηση πόρων θα μπορούσαμε να είχαμε. Επίσης, τονίσαμε τον αμέ της φορολόγησης της ρήπανσης. Η καινοτομία είναι ένα άλλο θέμα. Πρέπει να δούμε τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν για πολλούς από τους πόρους που σπανίζουν αυτή τη στιγμή. δεν μπορούμε να είμαστε τόσο εξαρτώμενοι από τις σπάνιες γέες όσο είμαστε τώρα. Και αυτό για να μπορούμε να έχουμε μια πολιτική περισσότερο ε, εστιασμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισχυρή στάση ε, που δείχνει ε, σε ορισμένους τομείς, γιατί πρέπει, οι πόροι, πρέπει τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν τη σημασία που έχει η αποτελεσματικότητα των πόρων. Και πρέπει τέλος να σκεφτούμε και τα θέματα των μοντέλων κατανάλωσης. Μακάρι να ήταν αρκετή η καινοτομία από μόνη της για να μπορέσουμε να έχουμε επαρκή αποτελεσματικότητα των πόρων στην Ευρώπη. Φοβούμαι ότι αυτό δεν είναι δυνατόν και πρέπει να μας απασχολήσουν και τα μοντέλα κατανάλωσης στην Ευρώπη και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα μοντέλα διατροφής μας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά συγκεκριμένα μέτρα και στον κατάλογο αυτό βλέπετε ε, ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι μια στρατηγική θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική μόνο όταν συμπεριλαμβάνει στοιχεία και από τις δύο πλευρές. Διότι βεβαίως πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία με καινοτομία, με ευελιξία, με εξασφάλιση του εφοδιασμού, αλλά θα πρέπει να τολμήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Πρέπει να φροντίσουμε να είναι οικολογικό ο σχεδιασμός των προϊόντων. Δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο στους εύκολους τομείς, θα πρέπει να κάνουμε ένα τολμηρό βήμα προς τα έξω και να μπούμε και σε τομείς που μερικές φορές δεν τολμάμε να αγγίξουμε. Και κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε στο μέσο μιας κρίσης ή στην αρχή μιας βιομηχανικής επανάστασης. Ούτως ή άλλως, ο επίγον χαρακτήρας είναι σαφής και πρέπει να δράσουμε γρηγορότερα από ό,τι τώρα, πιο γρήγορα από ό,τι κινούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το, και το Συμβούλιο των Υπουργών. Μία από τις βασικές προτεραιότητες, μία από τις βασικές ευθύνες του Κοινοβουλίου μας είναι να επιταχύνει τη διαδικασία μετάβασης προς ε, αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων στην Ευρώπη και περιμένω, κύριε Πρόεδρε, να ακούσω τις αντιδράσεις των συναδέλφων γιατί θέλω να τις συμπεριλάβω στο σχέδιο εκθεσής μου. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, thank you. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, ε, κύριε Γκέμπραντ, ε, για αυσιο έγγραφο που νομίζω ότι περιλαμβάνει πολλά καλά στοιχεία ε, για την, για την έκθεση που θα συντάξουμε αργότερα. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά εργαλεία και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και πολύ σωστά επίσης ε, αναφερθήκατε όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά και στους ε, καταναλωτές, στην κοινωνία που καλούνται να συνειδητοποιήσουν όλα αυτά και να μεταβούν ε, σε μια πιο σωστή συμπεριφορά κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους οι πολίτες. Έχουμε περίπου 20 λεπτά για συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιος άλλος επιθυμεί να λάβει το λόγο, γιατί προτίθεμαι να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Εσείς ε, προβλέπεστε, Γιούντι. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτούς που έχω στον κατάλογό μου. Ο Καλ Χάιντς Φλόρεντς ε, έχει βγει έξω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και ευχαριστώ τον συνάδελφο για αυτή την ε, θαυμάσια έκθεση και για τις ε, απόψεις σας. Και πρέπει να σας πω ότι σας στηρίζω στις δικές σας τις ε, φιλοδοξίες αλλά και αυτές της Επιτροπής. Και φαντάζομαι θα διαπιστώσετε ότι τα περισσότερα μέλη αυτής της Επιτροπής είναι εξίσου φιλόδοξα και στηρίζουν όλες αυτές τις απόψεις. Όπως είπαμε και στον Επίτροπο εξάλλου. Το θέμα όμως που τίθεται είναι πώς, πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Και αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία κατά πόσο μας προσφέρει αρκετά εργαλεία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να δουλέψουμε λιγάκι γιατί νομίζω ότι προφανώς ε, και όλοι θέλουμε να πετύχουμε ε, τα πράσινα λιβάδια και τον παράδεισο. Το θέμα είναι ο δρόμος που οδηγεί προς τα εκεί δεν είναι σαφής. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε ένα σύστημα ε, που θα επιτρέπει να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και αυτό να είναι το σύστημα που θα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν στην Ευρώπη κάποιοι πυρήνες ε, καινοτομιών, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών και ένα άλλο σύστημα που θέλω να αναφέρω. Κοιτάξτε, έχουμε τόσες πολλές ετικέτες, ε, οικολογικές, ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Στη τελική ανάλυση έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πλέον τι γίνεται με αυτές ε, τις ετικέτες, τα σήματα, το πράσινο η πράσινη, ο πράσινος κύκλος, παραδείγματος, γκρούνα πούντο, όπως λέγεται στα γερμανικά, κανείς δεν καταλάβαινε τι ακριβώς σήμαινε αυτό. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει κάποια διευκρίνηση, γιατί αυτή ε, θα καθορίσει και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η στάση των καταναλωτών είναι καθοριστική σημασία. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να την επηρεάσουμε. Και κάτι άλλο, ίσως οι πληροφορίες να μην αρκούν, να μην αρκούν οι ετικέτες. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα κίνητρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι είναι η καθήλυνα αρμόδια. Πρέπει να δούμε λιγάκι και το φορολογικό θέμα. Επίσης θα ήθελα να σας στηρίξω σε αυτό που αναφέρατε στο ότι ε, θα πρέπει να καταργηθούν οι ε, μη βιώσιμες ενισχύσεις. Αλλά και αυτό πάλι είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς θα το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να έχουμε μια γενική εικόνα της κατάστασης και μετά ενδεχομένως να καταργήσουμε αυτές τις επιδοτήσεις. Αλλά το θέμα είναι θα το κάνουμε με αυτήν την έκθεση ή μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να το παρακάμψουμε. Αναφερθήκατε στις καινοτομίες και εμείς βεβαίως το στηρίζουμε σε μία εβδομάδα. Η Κομισιόν θα έρθει με το μεγάλο πρόγραμμα, τον ορίζοντα του 2020, το μεγάλο αυτό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία. Και πιστεύω ότι αυτές οι απόψεις ε, που αναφέρθηκαν εδώ ταιριάζουν θαυμάσια στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και ελπίζω οι φιλοδοξίες μας να λάβουν πιο συγκεκριμένη μορφή. Πολύ ωραία, λέω. Πρόεδρος. Φαίνεται να κάνουμε λοιπόν πάρτι εμείς οι Ολλανδοί, οπότε ας τα πω τώρα και όχι αργότερα. Για την αποδοτικότητα και για την καινοτομία, γιατί αυτό μας αρέσει πολύ στους Ολλανδούς, μια και έχει προκλήσεις και ευκαιρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στο έγγραφό του και νομίζω πως έχεις όντως περιγράψει με άριστο τρόπο την κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι συγκεκριμένε προτάσει, τουλάχιστον από την πλευρά του Κοινοβουλίου, γιατί αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη μου ανησυχία. Δηλαδή, συμφωνούμε όλοι το πρόγραμμα και τη σημασία τη αποδοτικότητα στη χρήση των ενεργειακών πόρων και των υπόλοιπων πόρων και μετά το αφήνουμε στην τύχη του χωρί να το συνοδεύσουμε με συγκεκριμένε προτάσει. Εκεί λοιπόν πιστεύω πω η έκθεση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι πιο σαφή και να τονίζει προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση πως εάν θες να πάρεις τα θέματα αυτά στα σοβαρά, τότε θα πρέπει να επιταχύνεις, γιατί χρειαζόμαστε γρηγορότερους ρυθμούς από αυτούς που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους και φαίνεται και στο ε, έγγραφό σου Γιάνν, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποιους υποστόχους. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε πιο πολύ σε άλλα θέματα. Έχουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη χρήση γης και τη χρήση υλικών. Και οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να, προβλάβ, να προβλέπουν ολόκληρη την το βιομηχανικό κύκλο ζωής, ε, και τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και όχι μόνο την οικιακή χρήση, γιατί διαφορετικά στέλνουμε μισό μήνυμα. Και βεβαίως με τον τρόπο αυτό, αντί να λύνουμε το πρόβλημα, εξάγουμε το δικό μας αποτύπωμα του άνθρακα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στη χρήση των υλικών, στη χρήση υγιής, στη χρήση του νερού, ε, στα όσα θα πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν να δούμε και το θέμα της μετατόπισης του φορολογικού βάρους, γιατί αν εξετάσει κανείς την προϊστορία θα διαπιστώσει και το είπε και ο Επίτροπος, πως το κόστος εργασίας τα τελευταία χρόνια αυξάνεται 200% ενώ το κόστος των υλικών έχει αυξηθεί μόνο κατά 40%. Άρα λοιπόν ήταν πολύ λογικό η οικονομία μας να μην ασχολείται με το θέμα της μείωσης χρήσης των υλικών και απλώς προσπαθεί να μειώσει τη χρήση εργατικών χεριών. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια στιγμή με μεγάλη, με μεγάλη ενεργία και βεβαίως με μεγάλη εξάρτηση από την εισαγωγή υλικών. Εκεί λοιπόν θα βοηθούσε η μετατόπιση της φορολογίας, όχι λοιπόν φορολόγηση της εργασίας, αλλά φορολόγηση των υλών, των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και των υπόλοιπων υλικών. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσαμε εμείς να φέρουμε τη διαφορά. Χαιρετίζουμε λοιπόν την οδηγία αυτή η οποία θα ασχολείται με το θέμα της φορολόγησης των ε, πόρων γιατί θα δημιουργούσε αρκετή συζήτηση και ενδεχομένω θα κατέληγε σε συγκεκριμένε προτάσεις. Χαίρομαι που είσαι συγγετής, θα συνεργαστώ μαζί σου και νομίζω ότι είναι πολύ ε, συγκεκριμένη η δική μας άποψη θέλουμε και διάφορες κλαδικές ε, ε, προσεγγίσεις στο θέμα της γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής αλίας για την ε, χρήση και την ανακύκλωση των αποβλήτων από τους κλάδους αυτούς. Διαφορετικά, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, θα γίνει άλλη μια καλή έκθεση η οποία θα πεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ίσως για μία και μοναδική φορά συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο από τους ε, πράσινους. Ε, ε, στην πραγματικότητα οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί είναι υλοποιήσιμες. Η έκθεση του συναδέλφου είναι ένα σχέδιο εργασίας, είναι αν θέλετε η πρώτη προσέγγιση της έκθεσης που μας έστειλε η Επιτροπή και νομίζω η δουλειά που έχει γίνει είναι πολύ καλή. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα θέματα τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ε, υπάρχουν ε, δύο-τρία θέματα που θα επισημάνω για να μην μακρηγορήσω και βεβαίω μετά αν θέλετε μπορούμε να ξανασυζητήσουμε όταν θα μιλήσουμε για τι τροπολογίε. Όταν λοιπόν γίνεται λόγο ε, για την ενίσχυση των ε, εμπορικών στοιχείων των προϊόντων και λαμβάνοντα υπόψη την προστασία του περιβάλλοντο, θέλω να είμαστε πιο σαφεί. Θα το κάνουμε αυτό σε επίπεδο ευρωπαϊκό ή αναφερόμαστε εδώ σε προϊόντα που εισάγουμε. Παραδείγματο χάρη, προϊόντα που εισάγουμε από την Κίνα. Ε, θα ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα εργοστάσια που παράγουν διάφορα προϊόντα και θα πρέπει κανείς ε, να φοβάται για όλα αυτά που εισάγονται από την Κίνα. Εκεί εξάλλου όλα ε, καταλήγουν στις ε, χωματερές φίρδιν μίγδιν. Όλα μαζί. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια μόλυνση. Και τι θα κάνουμε με αυτά τα προϊόντα, θα τα αφήσουμε να μπαίνουν αυτά ανεξέλεγκτα στην Ευρώπη ή μήπως αγαπητέ συνάδελφε θέλετε να πευτείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τους πείτε, ξέρετε κάτι, αυτά είναι προϊόντα τα οποία έρχονται εδώ και μας μολύνουν, μας ρηπαίνουν. Ε, εφόσον μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία θα πρέπει να ισχύει για όλους, όχι μόνο για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Και μετά τι θα πούμε στην Επιτροπή, ξέρετε, ας προσπαθήσουμε να φορολογήσουμε αυτά που ρηπαίνουν και όχι τα άλλα τα οποία δεν ρηπαίνουν. Τι θα πούμε στην Επιτροπή, η οποία είναι εκείνη που εκπώνησε μία οδηγία στην οποία προβλέπεται απαγόρευση ε, φορολογίας ε, του ε, μεθανίου παραδείγματος χάρη ε, θα αυξήσουμε τα, τη φορολογία σε άλλα προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν εσείς να τοποθετηθείτε από αυτού. Δηλαδή, αν πρόκειται να φορολογούμε αυτό το οποίο ρηπαίνει, σε σχέση με το μεθάνιο θα πρέπει να φορολογήσουμε περισσότερο άλλες ρηπογόνες πηγές. Εξάλλου, θα πρέπει να δούμε και το εξή. Πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα εκείνα τα οποία οδηγούν σε μικρότερη ρήπανση. Τι μπορούμε να κάνουμε με ε, την, ε, τις μονάδες καύσης ε, που υπήρξαν κατά το παρελθόν και που θελήσαμε να κλείσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Όμως από εκεί κλείονται στην ατμόσφαιρα τα ε, σωματίδια και οι διοξίνες. Τι θα κάνουμε λοιπόν με όλα αυτά τα οποία χρηματοδοτήσαμε εν μέρει εμείς. Τι θα τους πούμε. Ξέρετε φίλοι μας ε, κάναμε λάθος και τώρα θέλουμε, ενώ σας χρηματοδοτήσαμε, τώρα θέλουμε να τα κλείσουμε. Κάτι πρέπει να πούμε για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να συνεργαστούμε για τέτοιου είδου θέματα. Και το τελευταίο που θέλω να πω και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι το θέμα ε, το PM10 και PM5, τα σωματίδια αυτά. Έχουμε τώρα κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ισχύουν για ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η Φινλανδία με 5 εκατομμύρια ε, κατοίκους ε, και με έκταση όμως ως Ιταλία ε, δεν μπορούν οι χώρες αυτές, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία που είναι εκβιομηχανισμένες να ανταγωνιστούν με άλλες περιοχές όπως η Φιλανδία που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη. γιατί μιλάμε για θέματα ε, τα οποία προσπαθούν να επιβληθούν σε χώρες όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Αν επιβάλλουμε αυτά τα όρια θα αναγκαστούμε να κλείσουμε βιομηχανίε στην Ευρώπη. Ας πούμε στην περιοχή Εμίλια Ρωμάνια. Εκεί μας λένε ότι για να παραμείνει κανείς μέσα στα όρια θα πρέπει να κλείσουν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες. Αρκεί ο αέρας να μεταφέρει την παραγωγή ε, από τη Λομπαρδία, από το Λάτσιο και φτάνουμε ήδη στα όρια. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να ε, εφαρμόσουμε κάτι το οποίο πραγματικά να είναι λειτουργικό πρόεδρος, δεν θέλουμε να κλείσουμε όλες τις παραγωγικές μονάδες. Εκείνο που θέλουμε είναι να τις αφήσουμε ανοιχτές, αλλά να μην είναι ρηπογόνες. Και ο τελευταίος ταρομιλητής, ο κύριος Σίμπα, πριν λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο σκιώδης ηγητής μας, ο κύριος Καρλ Χάιντς, δεν είναι εδώ ε, και γι' αυτό θα μιλήσω εγώ και εξ ονόματός του. Όταν μιλάμε λοιπόν για την αποτελεσματικότητα των πόρων, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον αφενός και αφετέρου να στηρίζουμε τη βιομηχανία. Γίνεται λόγος για αυτά τα περίφημα μηνύματα που έχουν σχέση με την τιμή. Ας μην ξεχνάμε ότι όσον αφορά τους πόρους ε, επαπειλείται η ε, έλλειψη. Υπάρχουν τομείς με μεγάλες αποτυχίες. Ανάλογο λοιπόν τώρα με το ποιος είναι ο στόχος, από εκεί εξαρτάται και η δομή τιμών που θέλουμε να επιβάλλουμε. Νομίζω αυτά είναι βασικά πολιτικά θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί νομίζω ότι υπάρχουν ε, ε, περιοχές ή τομείς αν θέλετε όπου ισχύει το θέμα των ε, τιμών και σε άλλους πάλι τομείς όχι το θέμα της καλής ατμοσφαιρικής ε, ποιότητας, ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, εκεί πράγματι τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αν δούμε λοιπόν τώρα αγαθά όπως είναι το νερό και ο καλός ατμοσφαιρικός αέρας, πρέπει να προσέξουμε να δούμε τι ε, περιοχές έχουμε στην Ευρώπη, γιατί επικύλουν κατά πολύ οι συνθήκες. Ας πούμε, σε μένα, στη δική μου την πατρίδα, ε, έχουμε επάρκεια υδάτριων πόρων. Και αν θέσουμε υπερβολικούς στόχους, κανείς δεν τους καταλάβει. Είναι αντιπαραγωγικό, σε τελική ανάλυση αυτό αντιβαίνει και στους στόχους. Αυτό δεν έχει άμεση σχέση με την καθαρότητα, ούτε με την οικολογική και χημική ποιότητα του νερού. Το να περιορίσει όμως κανείς το νερό στη χρήση του, αυτό έτσι και αλλιώ δεν φέρνει τίποτα, γιατί εξαρτάται στην περίπτωση αυτή κανείς περισσότερο από τους ποταμούς. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, τον οικολογικό σχεδιασμό. Αυτά πρέπει να δούμε κατά πόσον πράγματι ταιριάζει εδώ η αρχή, ένα μέγεθος ταιριάζει για όλα. Ε, εκείνο που θέλω να προβάλλω είναι το περιφερειακό στοιχείο. Οι περιφέρειες παίζουν ρόλο ε, και μην το ξεχνάμε γιατί χρειαζόμαστε και την αποδοχή των πολιτών. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για αποτελεσματικότητα των πόρων, θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς που κατευθυνόμεθα, να γνωρίζουμε τους μηχανισμούς που υφίστανται. Και να ξέρουμε κατά πόσον τα μέτρα ισχύουν για συγκεκριμένους τομείς, για το σύνολο των τομέων, μήπως ε, υπάρχουν περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Αυτό που παίζει ρόλο είναι οι αποχρώσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Όσον αφορά τους ε, γενικούς στόχους, νομίζω όλοι συμφωνούμε. Μόνο που η ε, δυσκολία βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Κατά την άποψή μου λοιπόν θεωρώ ότι είναι ε, πολύ μεγάλη επιτυχία της Κομισιόν αυτό το περίφημο mainstreaming, ε, δηλαδή περιφερειακή πολιτική, πολιτική ελίας, ε, πολιτική γεωργίας, το να αναγκαστούν αυτές οι πολιτικές και οι επίτροποι να λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία καθοριστικής σημασίας. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση και βεβαίως αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τον αρμόδιο επίτροπο. Πολύ ωραία. εκπρόσωπο της Γενικής διεύθυνση περιβάλλοντο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yeah, uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, εξαιρετική πρώτη παρουσίαση αυτής της εργασίας. Συμφωνούμε με αυτά τα οποία ως διάγνωση ανέφερε και συμφωνούμε με τις κατευθύνσεις τις οποίες ε, προανέφερε για την έκθεσή του. Και ευχαριστούμε και τους ομιλητές ε, για συγκεκριμένες υποδείξεις που έκαναν. Κύριε Γκέρβραντι, η Επιτροπή κατανοεί τον επίγοντα χαρακτήρα που και εσείς αναφέρατε και είναι αποφασισμένη να κινηθεί προς συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίηση όλων αυτών με την περαιτέρω επεξεργασία του οδικού χάρτη και περιμένουμε ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο το οποίο σιγά σιγά θα διαμορφώσει λεπτομερέστερα αυτές τις ε, ιδέες. Αυτή η έννοια του κατεπήγοντος ε, έχει ήδη ενταχθεί την ε, επιθυμία μας να έχουμε στόχους ε, μέχρι το 2013. Και ο τελευταίος ομιλητής ανέφερε πόσο σημαντική είναι η πρόκληση που τίθεται από τους ε, δείκτες τους οποίους θα παρουσιάσουμε. Αυτό τα γνωρίζει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για τους δείκτες που θα παρουσιάσουμε θα έχει γίνει ξεκάθαρη αξιολόγηση επιπτώσεων, επιπτώσεων στα κράτη-μέλη, σε διάφορους τομείς, όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Αυτό θα μας δώσει αποδεκτά αποτελέσματα τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας και περιμένουμε τη συνεργασία που θα έχουμε σε αυτό το δύσκολο τομέα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Επί δυόμιση ώρες μιλήσαμε για την αποτελεσματικότητα των πόρων, μια εξαιρετική συζήτηση, γιατί είναι και το θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Γκέβεν Γιάνν Γκεμπράντι άκουσε όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν και μέσα στην επόμενη χρονιά θα μας κάνει μια εξαιρετική έκθεση, την οποία θα συζητήσουμε και πάλι λεπτομερώς. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να σχολιάσει. Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γκερμπράντι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα σχόλια που άκουσα από τους συναδέλφους. Και η πολιτική μάχη θα αφορά αυτά τα οποία θα συζητηθούν για την φορολόγηση, την τιμολόγηση. Ε, και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, υπερβολικά σημαντικό για να παραμείνουμε κολλημένοι σε παλές ιδέες. Θέλω να διασφαλίσω και τον κύριο Αικάουτ ότι η έκθεσή μου θέλω να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ ε, για τα σχόλιά σα και για τη δουλειά σα και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι επίση ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο μέχρι το 2050. Και έχουμε τον Chris Davis ε, που είναι ο εισηγητή από του φιλελευθέρου, που μπορεί να μας παρουσιάσει τώρα την έκθεσή του. Chris Davis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δεσμευτεί ότι θα μειώσει τις εκπομπές μετά το 2020. Περιμένουμε μια διεθνή συμφωνία πριν περάσουμε σε υιοθέτηση πιο φιλόδοξων μέτρων. Τώρα πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε πιο, φιλόδοξα, πιο φιλόδοξη συμφωνία σε διεθνέ επίπεδο στο προσεχέ μέλλον. Ε, δεν τίθεται μόνο όμω το θέμα μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Ε, Περίπου το 12% των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εκπομπέ που οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά, αλλά δεν μπορούμε εμεί μόνοι μα να λύσουμε τα προβλήματα ολόκληρου του πλανήτη. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα στην οικονομία μα ε, και θα ήθελα να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα και να προωθήσουμε την οικονομία μας και να δώσουμε κατευθύνες γραμμές για τις επενδύσεις στο μέλλον. Αν δείτε τον ενεργειακό τομέα, η βασική προτεραιότητα για τις εταιρείες ε, ε, ενέργειας είναι το να ε, επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό οφείλεται στο ότι επιδοτούνται αυτοί οι τομείς από τις κυβερνήσεις. Τι κάνουμε όμως με τα ορυκτά καύσιμα. Αυτή τη στιγμή η τιμή για την το τίμημα για την ανάπτυξη των ορυκτών ε, καυσίμων ε, δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα μας επιτρέψει να κινηθούμε σε ένα ορίζοντα πάνω από 30-40 χρόνια. Κανείς δεν θα θέλει να επενδύσει σε κάτι και μετά από 40 χρόνια να έχει ε, στην διάθεσή του εξοπλισμό που θα είναι απερχαιωμένος ε, και πρέπει να δώσουμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές προς τους επενδυτές. Αυτός ο δικός χάρτης λοιπόν πρέπει να είναι κάτι που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω συγκεκριμένων προτάσεων για το μέλλον. Η έκθεσή μου είναι σύντομη Έχω τηρήσει τους ε, όρους ε, του Κοινοβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα του κειμένου και περιμένω ε, τις προτάσεις και τα σχόλιά σας για το κείμενό μου και πρέπει να πούμε ότι και η Επιτροπή Βιομηχανίας ψηφίζει αυτήν την εβδομάδα για την έκθεσή της. Όλες οι σχετικές συζητήσεις νομίζω βαίνουν προς την κατεύθυνση η οποία θα ήταν επιθυμητή και από την Επιτροπή μας. Τα βασικά στοιχεία τα οποία έχω στην έκθεσή μου είναι πρώτον να εγκρίνουμε τον οδικό χάρτη της Επιτροπής και τους στόχους ή ορόσημα τα οποία προτείνεται για το 2030 και το 2040. Και ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα θέσει τις βάσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε, να ρυθμίσουμε το θέμα των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος και το σύστημα εμπορίου εκπομπών. Είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, ε, το οποίο όμως ε, δεν καταφέρνει να προωθήσει επενδύσεις στον τομέα χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, πάντοτε υποθέταμε ότι μέχρι τώρα θα κόστιζαν τα δικαιώματα εκπομπών 30 ευρώ ανατόνο. Όμως, τα επίπεδα τα οποία τώρα βλέπουμε είναι πολύ πιο δυσμενή για την πολιτική την οποία θα θέλαμε να προωθήσουμε. Θέλουμε να κινηθούμε λοιπόν προς ε, μια κατεύθυνση μείωσης ε, των μακροπρόθεσμων εκπομπών και αυτή τη φορά μιλάμε ε, για μειώσεις 1,74% ετησίως για τα ανώτατα όρια Και για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους πρέπει να δώσουμε βεβαιότητα στους επενδυτές. Υπάρχουν κάποια αντιφατικά στοιχεία τα οποία θέλω να σας επισημάνω. Πρώτον, είναι το τρίτο στοιχείο το οποίο εγώ πρότεινα για να βελτιώσουμε το σύστημα εμπορίου εκπομπών, που είναι το να θέσουμε ένα, όριο, ένα ελάχιστο όριο για τη δημοπράτηση των συμβολέων των δικαιωμάτων εκπομπών. Δεν λέω ότι πρέπει να βάλουμε την τιμή ε, στο επίπεδο που θα θέλαμε να βρίσκεται, αλλά για να δώσουμε κάποια εμπιστοσύνη στους επενδυτές και να μην καταρρεύσει η αγορά, πρέπει να βάλουμε το όριο σε κάποιο σημείο όπου οι επενδυτές δεν θα φοβούνται ότι θα πάει εντελώ χαμένη η επένδυσή τους. Έχουμε κάνει τόση πολλή δουλειά στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και τώρα πια λυπάμαι, αλλά το σύστημα της εμπορίας εκπομπών δεν δίνει την βεβαιότητα που θα έπρεπε να δίνει στους επενδυτές. Ακόμη, η Επιτροπή πρέπει να θέσει τους νέους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 πρέπει να δούμε ποια είναι τα θετικά σημεία. Θέτουμε στόχους για να έχουμε σημαντικά επιτεύγματα. Να μειωθούν οι εκπομπές, να μειωθούν οι δαπάνες ε, του προϋπολογισμού μας. Αλλά αν θέσουμε ένα συγκεκριμένο στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές, τρευλώνουμε την αγορά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιτύχουν του στόχους μείωση των εκπομπών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις συγκεκριμένες δικές τους συνθήκες. Και αυτά είναι θέματα ανοιχτά προς και εγώ είμαι ανοιχτός προς συζήτηση. Πρέπει να δούμε αν λοιπόν είναι επαρκής και αν ε, εκπληρώνουν το στόχο τους οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Επιτροπή μας πολλές φορές έχουμε συζητήσει το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Η πυρηνική ενέργεια είναι ένας τρόπος για την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ορισμένα κράτη-μέλη θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να τους πούμε ότι αυτό αποκλείεται. Επίσης, όσον αφορά την δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν ε, να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία για την ε, αποθήκευση του άνθρακα ε, στο έδαφος. Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και αρκεί να διαβάσει κανείς τις εκθέσεις του Διεθνούς, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ε, που λέει ότι αν θέλουμε να μειώσουμε τους στόχους, ε, αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές και να φτάσουμε τους στόχους για το διοξείδιο του άνθρακος, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τον τομέα της ε, δέσμευσης και αποθήκευσης διοξείδιου του άνθρακα. Μία πρόταση που θέλω να υποβάλω εδώ σχετικά με αυτά τα οποία λέμε είναι ε, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα να έχουν άδεια λειτουργίας όχι παραπάνω από 10 χρόνια και στη συνέχεια να επανεξετάζεται η κατάστασή τους. Ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να πούν τα κράτη-μέλη ότι θα συνεχίσει να, να δουλεύει, θα συνεχίσει να λειτουργεί ε, αυτό το εργοστάσιο παραγωγής ε, ε, ενέργειας, εάν μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Δεν προσπαθώ να προωθήσω αυτή την πολιτική αυτή τη στιγμή, αυτή την τεχνολογία. Απλώς προσπαθώ να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις για να είναι εφικτή μια τέτοια πολιτική. Διαφορετικά υπάρχει ένας ε, πραγματικό κίνδυνος ε, ε, να καταφύγουμε στο φυσικό αέριο ως μόνη λύση μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική η οποία θα προωθεί τεχνολογίες ε, που στη συνέχεια θα πρέπει να, ε, να οδηγήσουν τους επενδυτές να κάνουν νέες επενδύσεις για να ε, εξοπλίσουν τα εργοστάσια τους με αυτά τα οποία θα απαιτούν οι τεχνολογίες της μελλοντική εποχής. Ένα επόμενο σημείο είναι η διαρροή διοξιδίου του άνθρακα, όπως αποκαλείται το να αγοράζουμε προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σε άλλες χώρες, οι οποίες εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα, δεν βελτιώνει την κατάσταση όσον αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήταν προτιμότερο να αγοράζουμε αυτά τα προϊόντα τα οποία θα έχουν παραχθεί στην Ευρώπη και θα, παράγουν θα εκπέμπουν το ίδιο διοξίδιο του άνθρακα. Και να αποφύγουμε λοιπόν την μετακίνηση της βιομηχανίας από την Ευρώπη σε άλλες χώρες λόγω της ε, πολιτικής μας για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι σημαίνει η προσαρμογή μας στην παγκόσμια οικονομία. Η παραγωγή αλουμινίου σαφώς έχουν πει ότι δεν υπάρχει μέλλον στην παραγωγή αλουμινίου πουθενά στην Ευρώπη. Βλέπουν εργοστάσια αλουμινίου να κατασκευάζονται ε, σε άλλα σημεία όπου υπάρχει φυσικό αέριο, παραδείγματο χάρη, στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα επιβολής ε, δασμών κατά την εισαγωγή προϊόντων τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε άλλες χώρες για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετεγκατάστασης βιομηχανιών ε, από την Ευρώπη σε άλλες χώρες. Ξεκίνησα τις παρατηρήσεις μου, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι σημαντικό είναι να δώσουμε ξεκάθαρες κατευθύνσεις στους Ευρωπαίους επενδυτές για να μπορέσουν να προωθήσουν ε, τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αν δούμε τι γίνεται στην Κίνα, τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, βλέπουμε ότι ε, κινούνται με πορεία ε, τέτοια που εμείς δεν μπορούμε ε, να παραμείνουμε σε απειχιωμένες τεχνικές. Αυτός ο δικός χάρτης ελπίζω, ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να κινηθούμε προς μια οικολογική κατεύθυνση, προς μια πράσινη κατεύθυνση που θα είναι η κατεύθυνση στην οποία θα ακολουθήσουν όλες οι προηγουμένες οικονομίες. Ελπίζω να μπορέσει και η Επιτροπή μας να συμφωνήσει και το Συμβούλιο το Μάρτιο να συμφωνήσει και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση εμείς προς το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Äh, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντέιβι. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για αυτή την ε, έκθεση η οποία περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία έτσι ώστε στα μέσα του αιώνα να μπορέσουμε να φτάσουμε σε βιομηχανικές μονάδες με περιορισμένες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η πολιτική εντυπωσιακό αυτό. Αποφασίζουν να χαράξουν ένα χάρτη πορείας για τα επόμενα 40 χρόνια. Και ε, από ό,τι φαίνεται το 2008, το 2009, πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, νομίζω ομόφωνα, δηλαδή και 27 αρχηγοί κρατών και, και κυβερνήσεων αποφάσισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 θα έχει μειώσει τις εκπομπές οξύτου του άνθρακα κατά 80 ή 90%. Δεν είμαι σίγουρος το κατά πόσον σήμερα αν αποφασίζαμε να λάβουμε αυτή την απόφαση θα το πετυχαίναμε. Πάντως έχει ληφθεί η απόφαση αυτή και κατόπιν τούτου είδαμε και στη στην προηγούμενη συζήτηση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων αναφέρθηκαν ε, αριθμοί όπως 7 δις σήμερα, 9 δις το 50. Όλοι λοιπόν επιθυμούν να έχουν ένα βιωτικό επίπεδο που θα είναι ικανοποιητικό και αυτό σημαίνει ότι αν συνεχίσει η χρήση των φυστάμενων πόρων αλλά και της ενέργειας θα πρέπει αναπόφευκτα να υπάρξει ένα είδο επανάστασης, βιομηχανική επανάστασης. Ελέγχθη αυτό και πρέπει να το επαναλάβουμε. Για αυτήν την έκθεση δεν είμαστε μόνοι μα. συνεργαζόμαστε με την έκθεση τη Επιτροπής βιομηχανία. Ο κύριος Περίλιο είναι ο εισηγητή τη Επιτροπής αυτή. Ε, δεν θα του δώσω τώρα το λόγο, θα του τον δώσω αργότερα. Το ανέφερα απλά και μόνο επειδή έρχεται από την Επιτροπή Βιομηχανίας και οι τροπολογίες που είδα εγώ είναι πάρα πολύ ικανοποιητικέ και γι' αυτό εάν περάσουν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε με ευρεία συνένεση σε πάρα πολλά θέματα. Εγώ λοιπόν είμαι σκιώδης ηγητής των σοσιαλιστών και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις το 80 μέχρι το 95% η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά αυτό το ποσοστό, αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει κατά 100% να είναι απελευθερωμένη, παντελώς απελευθερωμένη από διοξίδιο του άνθρακα. Ο κύριος Σεντέιβις ανέφερε μία σειρά δυνατοτήτων. Η ε, δυνατότητα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν τα εξή σενάρια ότι η Ευρώπη μέχρι το 2050 είναι αναμφίβολα σε θέση να ε, είναι αυτάρκη στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι άλλες εναλλακτικέ λύσεις, παραδείγματος χάρη η επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, αυτή είναι επίμαχη και ου αυτό, αλλά έχει και προβλήματα σε σχέση με τις επενδύσεις και την ασφάλεια. Η τρίτη εναλλακτική λύση η ε, περίφημη τεχνολογία CCS της αποθήκευσης και δέσμευσης του διευθύντου του άνθρακα και αυτή είναι ε, επίμαχη θα έλεγα. Ε, Πήγα, επισκέφτηκα την Ορβηγία, το Μόγκστατ, στη διάρκεια των προηγούμενων ε, διακοπών ε, του Πάσχα και εκεί έχουμε εταιρείε όπως την Alstom, την Ερβέ και πάρα πολλές άλλες πολυεθνικές που κάνουν δοκιμές. Πραγματικά σοκαρίστηκα εντυπωσιάστηκα από τις τεράστιες αυτές πολυεθνικές που κάνουν αυτές τις δοκιμές και θεωρώ ότι Ποτέ δεν είχα καταλάβει ότι χρειάζονται τόσο μεγάλες επενδύσεις για να καταργηθεί, για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μιλάμε δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα συνεπάγεται ένα τεράστιο κόστος. Κατόπιν τούτου στόχος μας θα πρέπει να είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 30, το 40 και μετά ίσως και το 50 όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση ενέργειας ε, προφανώς ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, η αποτελεσματικότητα της ενέργειας να είναι συνδυασμένη με την αποτελεσματικότητα των πόρων. Αυτό το σύστημα, το ETS ε, της εμπορίας εκπομπών δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο θα το επιθυμούσαμε. Όμως, ε, Κρίς, θυμάσαι, εδώ ήμασταν το βράδυ σε ένα δείπνο στο Κοινοβούλιο και ο κύριος Τεπέκια είπε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο της αγοράς και όταν δηλαδή υπάρχει ύφεση πέφτει η τιμή και όταν θα ανακάμψει η οικονομία θα αυξηθεί η τιμή. Πρέπει λοιπόν να δούμε λιγάκι πού ακριβώς ε, παρεμβαίνει η πολιτική. Ε, δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στον μηχανισμό της αγοράς, αλλά περισσότερο στο ότι εκδίδονται πάρα πολλά δωρεάν πιστοποιητικά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παρέμβουμε, ορισμένα εξ αυτών να τα απομακρύνουμε από την αγορά. Πάντως οι διακοιμάνσεις των τιμών, οι ανώτατες και οι κατώτατες ε, τιμές νομίζω ότι στρέφονται κατά αυτού του εργαλείου. Γιατί ούτε και η αγορά ίδια γνωρίζει πότε επέμβει την επόμενη φορά η πολιτική. Τι σημαίνει αυτό. Ένα εργαλείο της αγοράς πρέπει να μπορεί να λειτουργεί στην αγορά. Και όχι να χορηγούνται όλα αυτά ε, τα πιστοποιητικά, τα δωρεάν πιστοποιητικά. Αν αυξήσουμε τις ε, τιμές θα προκύψει ένα πρόβλημα που θέλω να το εξετάσουμε στην έκθεσή μας. Το πρόβλημα αυτό ε, είναι η ενεργοπαινία, η έλλειψη ενέργειας. Η πολιτική λοιπόν θα πρέπει να προσφέρει κάποια κίνητρα έτσι ώστε και οι φτωχότεροι πολίτες του πλανήτη να μπορούν ε, και αυτοί να συμμετέχουν στην ενεργειακή πολιτική. Όσον αφορά την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως, το είπατε κύριε Ντέιβις, η ε, βιομηχανία εξακολουθεί να έχει ε, μονάδες που παράγουν αλουμίνιο, χάλιβα. Εγώ στη δική εκλογική περιφέρεια έχω δύο μονάδες παραγωγής χάλιβα. Πρόκειται για μόνο παραγωγή ε, μονάδες που δουλεύουν με προϊόντα ε, που έχουν μία τιμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν είναι κανείς ε, πάνω ή κάτω αυτή την τιμή, θα πρέπει να δει πώς μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα του. Νομίζω ότι όλους μας ενδιαφέρει οι εταιρείε αυτές να μην μετεγκαθίστανται ούτε στη Μέση Ανατολή, ούτε να εξάγουν στην Κίνα, να μείνουν στην Ευρώπη. Βεβαίως για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες ε, κατά αυτών των μονάδων. Και εγώ στηρίζω το αίτημα προς την Κομισιόν να μας υποβάλει αναλύσεις, να μας δείξει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς τους τομείς και να δούμε πού μπορεί να βοηθήσει πολιτική. Ε, στην ενεργειακή πολιτική, στην κλιματική πολιτική. Να λάβουμε υπόψη μας αυτό το πρόβλημα της, ε, του ενδεχόμενου κατάσταση των επιχειρήσεων. Θέλω να σας πω ότι η βιομηχανία είναι ένας ε, σημαντικός τομέας, όμως το σύστημα των, της εμπορίας καλύπτει μόνο το 40% των ε, εκπομπών. Υπάρχουν και σε άλλους τομείς ε, εκπομπές ε, και αυτοί οι άλλοι τομείς πρέπει να καλύψουν το 60% γιατί αλλιώς δεν θα πετύχουμε τη μείωση κατά 85% ή 90%. Το τελευταίο που θέλω να πω αφορά στις εκπομπές που δεν έχουν σχέση με το διοξιδίο του άνθρακα. Το πρωτόκολλο του Μοντρέαλ στην έκθεση δεν αναφέρεται αναλυτικά εμείς εδώ εξετάσαμε το πρωτόκολλο του Μόντρελ. Αν ένα όχημα επηρεάζει ε, το κλίμα από 400 μέχρι 4.000 φορές, ε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αναφορά επ' αυτού. Ε, νομίζω ότι ε, μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά στο μέλλον. Ο κύριος Ζέμπα έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, μας δίνει το δικαίωμα να μιλήσουμε εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και εσείς ε, σκιώδης εισηγητής ε, και έχεις την ε, υποστήριξή μου και εγώ εκ μέρους της συναδέλφου λαμβάνω το λόγο. Θα ξεκινήσω με το σημείο στο οποίο ε, κατέληξες εσύ σχετικά ε, με τα αέρια εκπομπής. Ε, ίσως η Επιτροπή την επόμενη χρονιά μας προτείνει ένα face down αυτών των αερίων εκπομπών. Το 2050 το 40% θα είναι αυτά τα αέρια, τα φθοριούχα αέρια. Θα πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί για τα αέρια εκπομπών, ανεξάρτητα από το διοξίδιο του άνθρακα, και θα πρέπει να δούμε και τα θέματα κόστους. Μία γενική παρατήρηση. Ότι διάβασα ένα κείμενο ενό Αμερικανού επιστήμονα πολέμιου της αλλαγή του κλίματος σχετικά με την, το εμπόριο εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα ε, Όπου έλεγε ότι θα αποτύχει αυτό το σύστημα και αν δούμε τις τιμές για το διοξείδιο του άνθρακος. Νομίζω ότι βλέπουμε ότι καταραίει η αγορά των δικαιωμάτων, της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Αν εξελίσσονται κατά αυτόν τον τρόπο οι τιμές του διοξείδιου του άνθρακος, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί με τις τιμές που έχουμε ορίσει για το εμπόριο εκπομπών δεν μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε. θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες φιλοδοξίες όσον αφορά παγκοσμίω το εμπόριο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έχουν αυξηθεί κατά 5,3% οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα ε, παγκοσμίω. Αν συνεχίσουμε λοιπόν προ αυτήν την κατεύθυνση θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε να τηρήσουμε τους στόχους μας για το 2050 και δεν συμφωνώ απόλυτα με τη δική σου εκτίμηση. Ε, σχετικά με το κατά πόσο έπρεπε να τεθούν αυτοί οι στόχοι για το 2050 από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό το οποίο για μας είναι δεσμευτικό μέχρι τώρα είναι μόνο οι στόχοι για, τις, ε, ε, για το εμπόριο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε με συγκεκριμένα μέτρα να καταλήξουμε προς αυτή την κατεύθυνση της οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Είναι σωστό ε, εργαλείο το εμπόριο εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα ή πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο για να επηρεάσουμε την κατάσταση. Εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη και το ότι γίνεται πιο δαπανηρή η παραγωγή στην Ευρώπη έχει ως αποτέλεσμα αυτό το οποίο ονομάσαμε carbon leakage, δηλαδή τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών εκτός Ευρώπης. Ε, και αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Ε, πώς θα μπορούσε ε, να διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, τι θα μπορούσε να μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει νόημα να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα ε, όταν ε, αυτοί οι οποίοι εκπέμπουν ε, τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος δεν είναι πρόθυμοι να κινηθούν προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών. Από δικής μας πλευράς είναι σαφές ότι θέλουμε να κρατήσουμε το σύστημα του εμπορίου εκπομπών, δεν θέλουμε να έχουμε νέους δεσμευτικούς στόχους, αλλά θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί και πώς μπορούμε να το συνεχίσουμε για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και η ασφάλεια του προγραμματισμού είναι ένα βασικό στοιχείο η τεχνολογία που θα επικρατήσει δεν έχει τόση σημασία. Αν θα είναι η τεχνολογία CCS για τη δέσμευση και αποθήκευση διοκτήτου, αν θα κάνει κάτι άλλο, η αγορά θα το αποδείξει τελικά. Αλλά να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να μην τρέχουμε ε, προς τη μία την άλλη κατεύθυνση με βάση τα μηνύματα που παίρνουμε από τις επικρατούσες τιμές. Εμείς θέλουμε ε, να έχουμε ένα σύστημα ε, το οποίο να είναι λογικό και σε αυτό θα δώσουμε την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Και να με συγχωρεί ο συνάδελφος που του πήρα το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κρίς για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει. Ήταν πραγματικά πολύ δραστήριος και έκανε μια σειρά από εκδηλώσεις και ακροάσεις και πρέπει να πω πως εκπροσωπήθηκαν με πολύ δίκαιο και ισότιμο τρόπο όλες οι πλευρές. Αυτό που δεικνύει πως ο συγητής θέλει να συζητήσει το θέμα με όλους τους σκιώδεις συγητές και τον ευχαριστώ. Να σας πω πως η δική μου ομάδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και χαιρετίζει την ιδέα αυτού του οδικού χάρτη που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μείωση των εκπομπών αυτών των ε, ανθρακούχων ε, εκπομπών και ελπίζω πως αυτό θα βελτιώσει τις επιδόσεις μας, θα βελτιώσει το κλίμα εμπιστοσύνης και συμφωνώ και με το ε, ψήφισμα του Συμβουλίου που θα πρέπει τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν κάποιες μακροπρόθερμες στρατηγικές στο θέμα αυτό. Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις επιχειρήσεις, στις βιομηχανίες, σε όλους τους ενδιαφερόμενους και να τους πούμε πως μπορεί η καθυστέρηση στην εφαρμογή κάποιων μέτρων θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστο. Το 30% μέχρι το 2020, το, 60, το 40% μέχρι το 2030 και το 60% μέχρι το 2050 είναι οι στόχοι του οποίου μπορούμε να στηρίξουμε. Ε, μπορούμε να στηρίξουμε εάν βεβαίω υπάρξουν μερικές συμφωνίες ε, όπου βέβαια το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε το 10% των παγκοσμίων εκπομπών. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή μόνοι μα και διακινδυνεύουμε με να πλήξουμε την οικονομική ανταγωνιστικότητά μας εάν το κάνουμε μονομερός. Όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι και κυρίως ο Ρίτσαρτ και θα συμφωνήσω μαζί του απόλυτα, θα πρέπει να σταθούμε πολύ προσεκτικά στο θέμα των στόχων ή της νομοθεσίας που θα επιτρέψουν την διαρροή άνθρακα και την εξαγωγή θέσεων εργασίας σε άλλες χώρες. Ο Κρίς αναφέρθηκε ε, στον κλάδο του αλουμινίου επειδή μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής, την περασμένη εβδομάδα στην περιφέρεια μου ένας μεγάλος κατασκευαστής ανακοίνωσε πως θα κλείσει τις εγκαταστάσεις του και ένας από τους λόγους που εξήγησε αυτή την απόφαση ήταν το κόστος συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντολογικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο με εθνική νομοθεσία. Άρα λοιπόν χρειάζονται, χρειάζεται αλουμίνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα λοιπόν θα παράγεται αλλού και θα επανεισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλασικό παράδειγμα διαρροής άνθρακα. Κατανοώ λοιπόν την υποκρίση για το πώ οι υψηλέ τιμέ ενεργειακών προϊόντων δημιουργούν προβλήματα, άρα λοιπόν θα πρέπει εμεί να μην το επιτείνουμε ε, ε, επιβαρύνοντα με επιπλέον κόστο τι εταιρείε αυτέ. Μαζί με άλλου ευρωβουλευτέ από την περιοχή πάντοτε έχουμε ξεκαθαρίσει πω είναι πολύ δύσκολο να συμμορφώνεται κανεί με την νομοθεσία η οποία έχει συνταχθεί. Μπορεί λοιπόν στο μακροπρόθεσμο μέλλον ε, να φέρναμε κάποια αποτελέσματα, αυτό δεν είναι σίγουρο, αλλά σίγουρα αυτό που κάνουμε είναι βραχυπρόθεσμα να πλήττουμε την ανταγωνιστικότητα. Και χαίρομαι που ο Κρίς έχει εστιάσει την προσοχή του στο θέμα αυτό της διαρροής του άνθρακα, που είναι σημαντικότατο κατά τη γνώμη μου και δεν θα έλεγα πως υπερβάλλουμε, όπως λέει ο Κρίς. Νομίζω ότι συμβαίνει και υπάρχει και μία μακροπρόθεσμη τάση οι, βιομηχανίε οι βιομηχανίες εντατικής κατανάλωσης ενέργεια να φεύγουν από την Ευρώπη για τις προτάσεις του εισηγητή για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα θα έλεγα και πάλι να φανούμε συνετοί και να μην χαρτογραφήσουμε το ενεργειακό μείγμα του μέλλοντος βασιζόμενοι σε τεχνολογία η οποία ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς. Έχει τεράστιο δυναμικό, ναι, χρήζει περαιτέρω εξερεύνησης, ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν θα πρέπει να βασίζουμε την πολιτική μας επαναλαμβάνω σε τεχνολογία που δεν έχει δοκιμαστεί. Πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια βασική συνιστός αυτής της συζήτησης. Χαιρετίζω τα σχόλια του Κρίς. Νομίζω ότι είναι ένας αμαρτωλός ο οποίος τελικά πίστεψε. Είχαμε πει πως η πυρηνική ενέργεια θα αποτελέσει ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργειακού μας μείγματος και χαίρομαι που ο Κρίς συμφωνεί μαζί μου. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Βεβαίως έχουμε και τα γεγονότα στη Φουκουσίμα που μας οδηγούν στο να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την πτυχή της ασφάλειας, αλλά εφόσον λυθούν, νομίζω πως η πυρηνική ενέργεια θα αποτελεί μια βασική ενέργεια της ε, χαμηλής εκπομπή άνθρακα βιομηχανίας Ευρώπης. Καταγράφω για το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών, εμπορίας ανταλλαγών τι παρατηρήσει τους και βεβαίως πρέπει να διαμορφωθεί αν θα εξυπηρετήσει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Τώρα για την ε, νέα ζυγοστάθμιση αυτού νομίζω ότι θα πρέπει οι προτάσεις να μετρηθούν, να είναι επιτεύξιμες, βιώσιμες και να μην πλήξουν την οικονομική ανάκαμψη την οποία όλοι προσδοκούμε για την Ευρώπη. Και με αυτά να ευχαριστήσω τον Κρίς και ε, με χαρά περιμένω και τις επόμενες συζητήσεις που θα κάνω για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής Είμαι ο κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που όσοι είναι μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού στην Αγγλία συμφωνούν τόσο πολύ και στο κοινοβούλιο μας. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως οι συντηρητικοί πάντοτε χαίρονται όταν οι φιλελεύθεροι ε, μετακινούνται προς την κατεύθυνσή τους. Το αντίστροφο δεν τους ικανοποιεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι εσωτερικά θέματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι είναι η οικονομία της χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε απερίφραστα πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με την οικονομία μας και ο τρόπος που τα επιλύουμε γιατί όταν μιλάει για το IPCC κάποιος πράσινος όλοι γκρινιάζουν αλλά ξέρετε όταν ο Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια λέει πω πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Γιατί μέχρι το 2015 ε, ο προπολογισμό, ε, μάλλον οι δυνατότητε που έχουμε ε, για χρήση άνθρακα θα έχει θα έχει χρησιμοποιηθεί από τη βαριά βιομηχανία. Άρα λοιπόν αυτό το ανακοινοθέν τύπο ε, είναι ένα ανακοινοθέν που θα έπρεπε να το διαβάσουν οι συντηρητικοί στην Αγγλία γιατί μπορεί να τους δώσει κάποιες ιδέες και να μην επαναλαμβάνουν την καραμέλα του πυρηνικού. Ίσως δημιουργεί κάποια έκπληξη το γεγονός που συζητάμε και πάλι το μηχανισμό ανταλλαγής εκπομπών. Μας είπαν πως δεν πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα μέχρι να ξεκινήσει να τρέχει. Θα είμαι πολύ σαφής. Είμαι βέβαιος που μόλις ξεκινήσουμε, ο Ρίτσαρντ θα μου πει «Ε, μην το αλλάξουμε τώρα που τρέχει». Οπότε πάντα υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος να μην αλλάξουμε τίποτα ποτέ. Γιατί βέβαια γιατί να αλλάζει κανεί του κανόνε την ώρα που τρέχει το παιχνίδι. Αλλά αυτό θα μα το πείτε σε δύο χρόνια, είμαι σίγουρο. Πριν περάσετε λοιπόν στο επιχείρημα αυτό... Α, μάλιστα. Πριν λοιπόν χρησιμοποιήσετε, αυτό το επιχείρημα, κοιτάξτε τους κανόνες που δεν χρησιμοποιούμε σήμερα για το 2013. Γιατί 1η Ιανουαρίου του 2013, 2013 θα ξεκινήσουμε με την τρίτη φάση Μάθαμε πάρα πολλά μετά την πρώτη και τη δεύτερη φάση. Άρα λοιπόν ας χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα αυτά πριν μπούμε στην τρίτη φάση, δηλαδή πριν την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το 2020, γιατί διαφορετικά θα έχουμε τον οδικό χάρτη, όπου το 2005 θα φτάσουμε το 80%, το 40% το 2030, αλλά το 2020 θα είμαστε στο 20%. Μα αυτό είναι παράλογο. Και όλοι πρέπει να αναγνωρίζουμε πως αν, ξεκι... αν συμφωνείς με το 40% το 2030 και το 80% το 2050, τότε για ποιο λόγο να παραμείνει στο 20% για το 2020. Είναι παράλογο. Γνωρίζουμε επίση πω πολύ εύκολα μπορούμε να τα προσαρμόσουμε με πιο μεγάλη αποδοτικότητα στην ενέργεια, όπου εκεί δεν έχουμε παραδώσει τα υποσχόμενα και ελπίζω πως εκεί οι τροπολογίες μας θα ενισχύσουν το κείμενο γιατί αν δούμε μόνο το θέμα του eco-design δεν θα πάμε μακριά. Είναι υπερβολικά και καλυμμένο. Άρα θα πρέπει να το πούμε πιο ανοιχτά. Το σύστημα λοιπόν εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να αλλάξει πριν το 2013. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Με, την... με τον παροπλισμό Μιλάμε για διαρροή άνθρακα. Αλλά πηγαίνετε σε χαλιβουργίες. Εγώ πήγα στην Τάτα, στη χώρα μου. Αυτή τη στιγμή έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο παραγωγής χάλιβα. Και όταν τους ρώτησα γιατί, μας είπαν γιατί υπάρχει η πιθανότητα περιβαλλοντολογικών ε, νομοθεσιών που μας οδηγεί σε νέα τεχνολογία που έχει πολύ λιγότερες εκπομπές σε διοξίδιο του άνθρακα. Άρα λοιπόν αντί να εξετάζουμε μόνο τις απώλειες που συνοδεύουν αυτή την εισαγωγή νομοθεσίας, ας κοιτάξουμε και την καινοτομία την οποία μπορούμε εμείς μετά να πουλήσουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ε, χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που προσφέρει αυτή η νέα νομοθεσία. Να ένα επιχείρημα που κατερρύπτει τα επιχειρήματα των συντηρητικών. Θα ήθελα να πείσω τον Κρίς για το εξής. Αυτή τη στιγμή το CCS ε, που είναι η συμπαραγωγή ενέργειας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η συμπαραγωγή ενέργειας θα πρέπει να περιοριστεί στις βιομηχανικές διαδικασίες για τις οποίες είναι ο μοναδικός τρόπος μείωσης εκπομπών άνθρακα, για παράδειγμα στη Χαλιβουργία γιατί εκεί βέβαια χρειάζεται ο άνθρακας για να δεσμεύσει. Παρακαλώ να είστε πιο αποδοτικό στη χρήση του χρόνου ομιλία που έχετε, λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίω, Τότε στα γρήγορα να μιλήσω μόνο στο θέμα των εσόδων που θα έχουμε. Γιατί αν δείτε ποια θα είναι τα έσοδα από την σύστημα ανταλλαγή με εμπορίας ε, εκπομπών θα πρέπει τα έσοδα αυτά να χρηματοδοτήσουν την κατάλληλη τεχνολογία που θα είναι η τεχνολογία ε, που θα έχει χαμηλή χρήση διοξιδίου του άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό θα τις προωθήσουμε και θα, δώσουμε, θα δείξουμε το μήνυμα στον κλάδο πως δεν είμαστε εναντίον του, αλλά τον βοηθάμε να μετακινηθεί προς αυτή την οικονομία χαμηλών εκπημών σε άνθρακα που φαντάζομαι όλοι επιθυμούμε. Και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω να ήμουν αποδοτικός. Ναι, γιατί έχουμε καθυστερήσει, λέει ο Πρόεδρος, και έχουμε πολλούς. Ο κύριος Ρώση, παρακαλώ. Grazie Presidente. Beh, allora qui si... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ε, να γράψουμε μια τελείως ε, επιφανειακή έκθεση. Είναι σαν ε, να πλησιάζουμε το 2050 ενώ χτυπάω ξύλο βέβαια, το 2050 πολλοί από εμά δεν θα υπάρχουν ούτε σίγουρα όχι ως πολιτικοί, πόσο μάλλον να ζούμε κιόλας ως φυσική παρουσία. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα υπάρξουν ε, λοιπόν κάποια συγκεκριμένα όρια. Είναι δύσκολο να ορίσουν τώρα. Μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα και για νέε δεσμεύσει, που βεβαίω και είναι αυτό ευκταίο. Όμω ε, εμεί το επιθυμούμε κάτω από το πρίσμα ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα βιομηχανισμένα κράτη. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν δυστυχώ πολύ στηρίζουν μία ένα μονόδρομο, ενώ από την άλλη, όπως σας είπα, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Κατόπιν τούτου, ελπίζω να έχουμε ακόμα εδώ έναν εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Ε, δεν ξέρω, ο πρόεδρος θα μας πει, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς πιστεύει η Κομισιόν σχετικά, ε, έστω και με τη μονομερή δέσμευση της Ευρώπης. Μετά υπάρχουν θέματα που με ανησυχούν, παραδείγματος χάνει. δέσμευση του Άντρακα. Ε, η εξάντληση των κοιτασμάτων, ορισμένων κοιτασμάτων. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τέτοιου είδους ε, προβλήματα. Με απασχολεί πάρα πολύ η δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα γιατί δεν θα ήθελα να συμβεί ε, κανένα ε, σοβαρό ατύχημα το οποίο θα έθετε σε κυκλοφορία αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι συγκαλυμμένα αλλά και άλλες επικίνδυνες ουσίες. Εξάλλου μας ανισχύει πάρα πολύ το θέμα του ντάμπινγκ γιατί με τον τρόπο αυτό η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει, θα αντιμετώπιζε ακόμα πιο πολλά προβλήματα. Ντάμπινγκ, ε, αθέμητος ανταγωνισμός από τις ε, τρίτες χώρες. Αυτό μας απασχολεί πολύ. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε σε όλα τα έγγραφα που φεύγουν από το Κοινοβούλιο να εντάξουμε και αυτή μια τέτοια πρόταση που να απαγορεύει το οικολογικό dumping όχι μόνο σε μονάδες που παράγουν αλλά και σε πολύ μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή και χαίρομαι που λέει ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ποιες ε, είναι οι κίνδυνοι της μετεγκατάστασης και ο πρόεδρος ε, κύριος ε, Λάιμπνεν είπε ότι ήταν καλό η Κομισιόν να μας ε, ενημερώσει για τους κινδύνους που υπάρχουν και συμφωνώ επίση με τον εισηγητή όσον αφορά τους δασμούς. Βέβαια, το θέμα των δασμών, των εισφορών, των δασμών από τρίτες χώρες που ε, δεν ε, σέβονται τους δικούς μας τους ε, κανισμούς. Ελέγχθη αυτό, αλλά πρέπει να είναι και σε γραπτή μορφή, γιατί νομίζω ότι με τρόπο αυτό θα βελτιωνόταν η κατάσταση. Επίσης, είναι σημαντικό να ορίσουμε και τις ποσότητες και το κόστος, την τιμή ε, του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί αλλιώς ε, υπάρχει κίνδυνος υπερεκμετάλλευσης ε, των, του συστήματος ανταλλαγών. Θα περάσω πολύ γρήγορα σε αυτό το σχέδιο του κυρίου Ντέβης, κυρίως σε αυτό το σημείο που προσπαθεί να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε ιδίως αυτό τον κίνδυνο της μετεγκατάστασης. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την διάταξη και θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τον εισηγητή να επανέλθει στο θέμα των δασμών γιατί νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να εισπράξουμε χρήματα έτσι ώστε να επιφέρουμε μία αντιστάθμιση. Δίνουμε το λόγο τώρα στους επόμενους ομιλητές, δύο λεπτά όμως, όχι παραπάνω. Πέτερ Λίζε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Κρις Ντέιβις για το σχέδιο έκθεσης. Είναι σημαντικό το ότι πρέπει να δώσουμε μακροπρόθεσμες προοπτικές για τη βιομηχανία και να δείξουμε σαφώς ότι θέλουμε να συνεχίσουμε και μετά το 2020. Εγώ πιστεύω ότι η στόχη του 2030 είναι πιο σημαντική και δεν αργεί να φτάσει το 2030 θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουμε να περιγράψουμε τους στόχους μας για περισσότερο μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά την τιμή του διοξιδίου του άνθρακα, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί είναι πρόβλημα όχι μόνο για τις επενδύσεις, όταν είναι συνεχώς χαμηλή η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και έχουμε προγραμματίσει και τα έσοδα από το διοξίδιο του άνθρακος για να επιτύχουμε τους στόχους μας και στη Γερμανία είναι σαφές αυτό όταν υπολογίζουμε ε, τις επενδύσεις που χρειάζονται και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν δεν υπάρχουν έσοδα, καταραίει ολόκληρη η στρατηγική μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή, εάν ε, έχει κάτι ε, για, να μας πει για, το, για τις τιμές του διοξιδίου του άνθρακα μετά το 2030. Τώρα είναι φθηνά τα δικαιώματα εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Θα συνεχίσουν να είναι και στο μέλλον, θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Ποια είναι η προοπτική. Το θέμα της διαρροής άνθρακα, του carbon leakage, για τη την των βιομηχανιών εκτός Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα πρέπει να τεθεί ένα στόχος πάλι και για το 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του προγραμματισμού το να έχουμε τέτοιους στόχους. Ευχαριστώ τον Chris Davis που χρησιμοποίησε πάρα πολύ αποδοτικά τις δυνατότητες που του δίνει και η Επιτροπή Ήτρε. Ε, ευχαριστώ και την ε, ε, γραμματεία και νομίζω ότι πολλά πράγματα θα πρέπει να συνεχίσουν να τα εξασφαλίζουν οι γραμματείες των Επιτροπών στη συνεργασία. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Πιερίλο, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ενημερώσω τους ε, συναδέλφους ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, για τον χάρτη πορείας ε, θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Εμείς κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Θα υπάρξουν 11 συμβαστικές προτάσεις που συγκεντρώνουν πάνω από 100 τροπολογίες και η Επιτροπή Βιομηχανίας με βάση το άρθρο 50 του κανονισμού ε, τελικά καταλήγει στο ότι ε, έχουμε θετικό αποτέλεσμα και ελπίζουμε σε αυτό να συγκεντρώσουμε τη τη δυνατή πλειοψηφία. Η έκθεση του συναδέλφου κυρίου Ντέιβις για μένα είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα κράτη-μέλη ε, πρέπει πράγματι να καταρτήσουν ε, το κάθε ένα από αυτά το δικό του χάρτη πορείας. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας το πρόγραμμα, θέλω να πω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς ε, για να κάνουμε μία σε ε, εκτίμηση του αποτελέσματος των επιπτώσεων ε, του συστήματος των εκπομπών. Πρέπει να εξετάσουμε το γεγονός ότι η τιμή ανατόνου διοξιδίου του άνθρακα έχει πέσει και για τις ε, βιομηχανίες ε, αυτή τη στιγμή ε, είναι πολύ πιο οικονομικό να συνεχίσουν να παράγουν με το ισχύον σύστημα και όχι να επενδύσουν σε μελλοντική τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν καλείται να κάνει εντελεχή ανάλυση σε πολλούς τομείς και για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να περάσουμε στην τρίτη φάση εφαρμογής του συστήματος ανταλλαγής αλλά ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις όλου αυτού του συστήματος. Επόμενος ομιλητής, κυρία Γκουτιέρες, ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως είναι πολύ γενικόλογο αυτό που θα πω, αλλά σημαίνει κάτι σε όλα τα έγγραφα και δεν θέλω βέβαια εγώ να καταρρύψω αυτούς τους πόθους και τις ελπίδες των συναδέλφων, αλλά για το 2020-2030 για τη μείωση των εκπομπών με εκπλήσει αυτό το πνεύμα βιωσιμότητας το οποίο υποτίθεται πως θα συγκρίνει μεταξύ τους τις επιπτώσεις της νομοθεσίας με το πλήγμα που θα φέρει έχουν μείνει τελείως εκτός συζήτησης γιατί με τον τρόπο αυτό συντάσσουμε οδηγίες οι οποίες μετά δεν εφαρμόζονται καταπληκτική νομοθεσία για βελτίωση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Αλλά δυστυχώς μένουν εκτός πεδίου, που είναι η δική μας οδηγία, που είναι η μείωση των εκπομπών στη βιομηχανία. Κάποια φορά θα πρέπει να συζητήσουμε ε, όλους τους κλάδους στους οποίους γίνεται αυτή η μελέτη του pre-impact. Γιατί επειδή πολλοί από εμά ζούμε σε χώρες σε κρίση, το να στηρίξουμε οι πολιτικές οι οποίες θα μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τις εκπομπές μας ζητάτε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει λόγο να γίνει. Είναι ασύμετρη η απειλή. Είπαμε στην αρχή βιομηχανία και αυτοκίνητα. Τώρα μιλάμε για τα κτίρια, για την αναβάθμιση των κτιρίων, την ενεργειακή. Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ίσως εκεί θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε χώρους πρασίνου στις πόλεις μας, στα σπίτια μας. Γιατί, και κλείνω τώρα, θα μπορούσε να αυξήσει την εξοικονόμηση αυτή με εντυπωσιακό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και ποιος είναι ο κατάλογο επιχειρήσεων όπως η Arcelor που φύγανε από την Ευρώπη για να πάνε κάπου αλλού να παράγουν, ε, να παράγουν ε, μια και υπάρχουν κράτη πολύ πιο φθηνά, ε, με λιγότερη νομοθεσία. Άρα λοιπόν παρακαλώ η αντιμετώπιση του θέματος να είναι σφαιρική. Έχω σημειώσει τους ομιλητές, ε, θα σας δώσω και σε άλλους τον λόγο, εάν παραμείνετε όμως στον χρόνο που σας έχω δώσει. Σάτου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Μιλάμε για μία μακροπρόθεσμη πρόπτικη, την οποία θα πρέπει μέχρι το 2050 να εφαρμόσουμε σιγά-σιγά, για να μπορούμε να πούμε ότι δεν θα αποτύχει αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα βοηθήσουμε τους κλάδους της βιομηχανίας ήδη από σήμερα. για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να υπολογίσουν πώς ε, θα οργανωθούν για να επενδύσουν στη σύγχρονη τεχνολογία. Και για το σύστημα των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσει τον εξυγχρονισμό της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση στο οποίο το επιθυμούμε. Η έκθεση του Chris Davis μιλά και για τις νέες τεχνολογίες και αυτό είναι σημαντικό γιατί πρέπει να τονίσουμε ε, τις επενδύσεις στην καινοτομία και στην έρευνα. Αυτό θα δώσει τη σωστή όθηση γιατί η βιομηχανία θα προσπαθήσει να επενδύσει εκεί όπου υπάρχουν υψηλότερε επενδύσει. Η κυρία Χίμπνερ ήταν η ομιλήτρια και τώρα η επόμενη ομιλήτρια είναι η Σάτου. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που καθυστέρησα, καθυστέρησε η πτήση μου όμως. Το πιο σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή εισήγηση. Συμφωνώ με τη βασική ιδέα ότι πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουμε με την πρόταση της Επιτροπής για τον Οδικό Χάρτη για το 2050. Όμως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σχέδιο της έκθεσης, μου άρεσε πολύ μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια να τεθεί ένα όριο 100 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακος ανά κιλοβατόρα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και κρίμα που δεν είχε αναφερθεί και στο παρελθόν όταν υπήρχε σχετική νομοθεσία, όπου θα υπήρχε δυνατότητα να προωθήσουμε αυτή την πολιτική. δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χάρτης πορείας της Επιτροπής ναι μεν είναι αρκετά φιλόδοξος ούτως ώστε να τηρήσουμε τους στόχους μας για την πολιτική του κλίματος, αλλά δεν είναι αρκετά φιλόδοξος για την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώνω τη συζήτηση και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 6 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα την ακούσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά ο κύριος Βιβάν περιμένει δύο ώρες τώρα. Δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε μετά το επόμενο θέμα. Ξέρω, λυπάμαι, θα έπρεπε να ακούσουμε την Επιτροπή. Μα... Μα δεν είναι αποδεκτό αυτό, λέει ο κύριο Κρι Ντέιβι. Να το αφήσουμε για αύριο το πρωί, αν δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Από ό,τι μου είπα, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, λέει ο πρόεδρο. Δεν μπορούμε να μην δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει έρθει εδώ ο υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει το χρόνο. Δεν μπορούμε να μην του δώσουμε το λόγο. Δώσω μόνο ένα λεπτό στην Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό, λέει ο κ θα πρέπει να το συζητήσετε και με τον ε, γιο τότε, με τον Γιώ Επιτροπή. Ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο, θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ τον εισηγητή, πολύ ισορροπημένη έκθεση που παίρνει υπόψη της και τα τρία βασικά που είναι και η ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και μας δίνει και κάποιες ε, προτάσεις για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς τα επόμενα τρία χρόνια. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που έχετε πει και για τα 2020 και για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τους χλωροφθοροάνθρακες, όλα αυτά βρίσκονται στο πρόγραμμά μας, άρα λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντικό το σχέδιο έκθεσης να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να προσπαθήσει να το επιλύσει. Αυτό έχει σημασία και για το βιομηχανικό μας κλάδο, γιατί χρειάζεται να έχει μακροπρόθεσμη βεβαιότητα για να κάνει τις κατάλληλες επενδύσεις στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τη διαρροή άνθρακα και όταν φτάσουμε αυτά τα ορόσημα θα πρέπει να τις ημερομηνίες αυτές θα πρέπει να δούμε πώς ε, δεν θα πλήξουμε ε, τις βιομηχανίες μας. Για τη συμπαραγωγή ενέργειας καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον εισηγητή και για τη χρονική στιγμή που το καταθέτει να σας πω πως εμείς είμαστε στην ώρα μας. δηλαδή για, τις, ε, για την, ε, ε, όλες τις προσπάθειες που έχετε περιγράψει δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχουμε τις αποφάσεις μας στα τέλη του 2012. Και πρέπει να σας πω πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και από πλευράς μας έτσι ώστε να έχουμε και κάποια μοντέλα τα οποία θα τρέξουν για να μπορέσουμε να κάνουμε εκεί τις δοκιμές. Ευχαριστώ. Και το 50% λοιπόν ήταν πολύ γενναιόδωρο. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο και λυπάμαι που περιμένατε τόση ώρα κύριε Ζουβά. Σας παρακαλώ πολύ έχετε το λόγο. Είναι για τους κινδύνους που προέρχονται από φυσικούς παράγοντες και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ευχαριστώ πολύ. Όχι μόνο εγώ, αλλά ε, και οι συνάδελφοι και οι σκιώδες και η κυρία Μωρά Σαχτιέ ε, την οποία ορίζουμε που είναι και η συγγήτρια στην Επιτροπή Απασχόλησης. Λοιπόν, το 2004 είχαμε μια οδηγία η οποία ήθελε να ορίσει κάποιες ανώτατες τιμές ε, αυτές τις ε, εκπομπές για τις μαγνητικές τομογραφίες που βοηθούν πάρα πολύ τη διάγνωση και τη θεραπεία κάποιων ασθενειών και φάνηκε πως αυτά τα ανώτατα όρια έκθεσης στο κείμενο από τον ιατρικό κόσμο θεωρήθηκαν δυσανάλογες γιατί δεν επιτρέπουν την ικανοποιητική διεξαγωγή αυτών των ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες ε, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές και για την καρδιολογία και για την νευρολογία και για την αγκιολογία και εκεί πραγματικά θεωρείται ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Λύνουν πάρα πολλές παθολογικές καταστάσεις και είναι πάρα πολύ, ε, πάρα οι καρκίνοι, όπως επίσης και οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες, οι οποίες χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εξετάσεις. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο κείμενο, το οποίο θα επέτρεπε να εισάγουμε και νέες ανώτατες τιμές για την έκθεση, καλό αυτό, για τις ιατρικές εξετάσεις, αλλά επίσης κάποιες εξαιρέσεις για ιατρικό εξοπλισμό ε, σε περίπτωση που έχουμε τέτοιου είδους μαγνητικές τομογραφίες, δηλαδή να στηρίξουν τους κανόνες εξαίρεσης, αυτό προτείνω και εγώ, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που ε, χειρίζονται τα μηχανήματα αυτά να μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν τις εξαιρέσεις αυτές. Είναι το τέλος σήμερα σήμερα αυτές οι εξαιρέσεις. Αν δεν γίνουν δεκτές νομίζω πως τελικά ε, ένας ολόκληρος κλάδος ε, εργαζομένων στον ιατρικό χώρο θα καταρρεύσει. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. Merci and thank you for... Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω με τους και Μουρίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που άφησες να γίνει αυτή η συζήτηση. Κρίμα που περιμέναμε τόση ώρα. Συγχαρητήρια στον κύριο Ζουβά, εξαιρετική η γνωμοδότηση. Το, μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι το ε, στηρίζω, πολύ πιο σαφές από τις προτάσεις της Κομισιόν και πολύ σωστά εστιάζει στην εξαίρεση για τη χρήση των τομογράφων, γιατί θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των πλεονεκτημάτων για τη δημόσια υγεία και των αρνητικών ε, συνεπειών για τους εργαζομένους που τα χειρίζονται. Προφανώς χρειάζονται οι τομογράφοι να εξαιρούνται από την νομοθεσία γιατί είναι πιο ασφαλής ε, και η μόνη εναλλακτική είναι ε, είναι βέβαια η χρήση ακτινογραφίας που είναι καρκινογόνος ενδεχομένως. Χρησιμοποιούνται για πάρα πολλές ασθένειες και αυτή τη στιγμή γίνεται και έρευνα για νέα χρήση των τομογράφων. Δεν είναι εύκολο να ε, εξασφαλίζουν πως είναι μακριά από τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται ε, από τους ε, ασθενείς γιατί τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται βοήθεια μέσα στο μηχάνημα και βέβαια ε, χρησιμοποιούνται τομογράφοι και κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων, άρα λοιπόν πρέπει να είναι κοντά στο πεδίο τους η, ε, το προσωπικό του χειρουργείου. Συμφωνώ με την εξαίρεση, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να μην ε, υποβάλουμε σε αυτό το προσωπικό σε διακρίσεις. Γι' αυτό το νέο άρθρο αυτό για τις εξαιρέσεις με βρίσκει λίγο διστακτική. Πιστεύω πως ίσως έτσι ανοίγουμε το ένα παραθυράκι έτσι ώστε άλλοι εργοδότες από άλλους κλάδους που θα ζητήσουν εξαιρέσεις να βασιστούν σε αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πως η εξαίρεση αυτή είναι ειδική περίπτωση και θα πρέπει να έχει και μια ενσωματωμένη ρήτρα αναθεώρηση έτσι ώστε να το ξαναεξετάσουμε. Θα πρέπει να δούμε πως παρόλο που οι χειριστές τομογράφων αποκλείονται από τα ανώτατα όρια, καλύπτονται από την οδηγία για όλο τον προστατευτικό, για την προστατευτική νομοθεσία. Και χαίρομαι που ο κύριος Ζουβά θα διαγράψει τους ξεχωριστούς ορισμούς ε, των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και ε, το θέμα για την προστασία. Προφανώς οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια για την, υγεία, για την υγεία θα ε, θίξει και την ασφάλεια του εργαζομένου και το αντίστροφο. Έχουμε διαφορετικά ανώτατα όρια έκθεσης και ε, για την υγεία και για την ασφάλεια. Άρα εκεί νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια λόγη Θέλω κάποιες διευκρινήσεις για την πρόταση να συνδυάσουμε τον ορισμό για την άμεση και έμεση, άμεσες και αρνητικές συνέπειες, μια και ε, κατανοώ για ποιο λόγο η Κομισιόν τα χώρισε μεταξύ τους. Και τέλος, παρόλο που έχει αφήσει εκτός τη ορετική δράση σε αυτών των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εκτός, γιατί δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία, θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι, γιατί εάν έχουμε κάποιες ιατρικές πληροφορίες για το θέμα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν αμέσως, αμέσως υπόψη για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Η αρχή της πρόληψης για να προστατεύσουμε τους χιλιάδες εργαζομένους που εκτίθονται σε τέτοια ηλεκτρομαγνητικά πεδία κάθε μέρα από τον κίνδυνο των σωρευτικ, της σωρευτικής έκθεσης. Ευχαριστώ τον κύριο Ζουβέν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή από, για την έκθεση από την Επιτροπή Απασχόλησης και νομίζω βιάστηκα όσο μπορούσα. Thank you. Ε, Γιάννα Κοντάκη, next. Γιάννα Κουδάκη, παρακαλώ. Και εγώ θα βιαστώ, θα μιλήσω γρήγορα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την πολύ καλή δουλειά. Ε, κατόρθωσε να επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στο να κατανοήσουμε τα ιατρικά ωφέλη και να υπάρχει επίσης ισορροπία με την ασφάλεια των ε, αξονικών τομογράφων. Είναι πολύ σημαντικό ε, να γνωρίζουμε ότι το κείμενο της Κομισιόν πρέπει να διευκρινιστεί. Επίσης, ε, ε, θα ήθελα να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, να μην είμαστε ιδιαίτερα περιγραφικοί στο να ορίσουμε ε, τους, ε, τις εξαιρέσεις και τις ε, αποκλήσεις. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τους μαγνητικούς τομογράφους νομίζω ότι η απάντησή μας θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογη με, τις, με τους κινδύνους. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξή. Μιλήσαμε για τη χρήση των μαγνητικών τομογράφων για λόγους υγείας. Πρέπει να ζητήσουμε εξαίρεση για λόγους έρευνας και επιστημονικούς. Πολύ καλή δουλειά ε, και πολύ καλή δουλειά και του εισηγητή ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Ο επόμενος είναι ο κύριος ε, Γιάννος Άντε. Δεν θέλω τώρα να διαβάσω αυτά που έχω γράψει. Θα ήθελα απλά να πω στους συναδέλφους που είναι παρόντες να απευθυνθώ στο συνέστημά σας. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά είμαι δυνάμι ασθενής. Και γι' αυτό λοιπόν έχω άποψη για το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 7 χρόνια έκανε ένα λάθος, υπέπεσε σε ένα σφάλμα. Μάλιστα αυτό αποτελεί σκάνδαλο, σκάνδαλο το γεγονός ότι δεν έφτασαν 7 χρόνια για να επανορθώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιο είναι το λάθος αυτό. Είναι ότι περίπου ένα πέμπτο των ασθενών, μάλλον κάθε πέμπτος ασθενής, στον οποίο χρησιμοποιείται μαγνητικός τομογράφος, επαναλαμβάνω, κάθε πέμπτος ασθενής που εξετάζεται με τη χρήση μαγνητικού τομογράφου, δεν μπορεί πλέον να έχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό είναι απαράδεικτο. Οι ε, γιατροί το είπαν πριν από αρκετά χρόνια, ήδη το 2001, ότι αυτή η ρύθμιση είναι απαράδεικτη και το νοσηλευτικό προσωπικό είπε επίσης ότι δεν υπάρχουν ε, βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία, στη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Και τώρα έχουν περάσει Επτά ολόκληρα χρόνια και αντί να λέμε την αλήθεια, εξακολουθούμε να συζητάμε για λεπτομέρειες. Οι συνάδελφοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει διάσταση απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ευσταθεί και η άποψη της ε, Επιτροπής. Όμως ε, πρέπει να πούμε ότι στο Συμβούλιο υπάρχει μια μειοψηφία που αποτελείται από 7 κράτη, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Λιτουανία και Τσεχία. Αυτές οι 7 χώρες πρέπει να πιστούν για το ότι ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει είναι το λιγότερο θα έλεγα ολιστηρός. Και δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο είναι ο ε, υπέτειο αυτού του σφάλματο. πρέπει λοιπόν να επανορθωθεί και στο μέλλον θα πρέπει η σύγχρονη αυτή τεχνολογία ε, να προσφέρεται σε όλους τους ασθενεί. Εσείς δεν είστε στον κατάλογο ε, για του σκιώδει, αλλά πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει κυρία Περβανόβα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει για το κείμενο αυτό. Ε, η ομάδα μας υποστηρίζει την προσέγγιση του και επίσης ε, εκτιμούμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα για τους μαγνητικούς ε, τομογράφους δίνοντας αυτή την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής. Και η συνάδελφος Φρεντερή Κρίστ το Φεβρουάριο του 2009 ε, πρότεινε παρόμοια μέτρα και είναι πολύ πλοκό και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο να διορθώσουν σφάλματα του παρελθόντος. Ελπίζουμε ότι δεν θα, ε, δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον αντίστοιχα σφάλματα. Έχει δοθεί λοιπόν αυτή η εξαίρεση όσον αφορά ε, τους κινδύνους για τους εργαζομένους. Βέβαια, ε, μια εξαίρεση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και πάντοτε φροντίζουμε να υπάρχουν τα επαρκή μέτρα ασφαλείας και προστασίας για τους εργαζομένους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων που έχουν σχέση με διαδικασίες σχετικά με μαγνητικούς ε, τομογράφους. Υπάρχουν ε, τα θέματα της μακροπρόθεσμης έκθεσης σε μαγνητική εκνοβολία από τη χρήση παραδείγματο χάρη κινητών τηλεφώνων. Αυτό είναι διαφορετικό πεδίο στο οποίο ε, απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή και πάλι. Ε, η συγγήτρια κυρία Μοχάν Σαχτιέ ε, ως συγγήτρια από την ε, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Ζουβάν και να τονίσω και εγώ τον επίγοντα χαρακτήρα που τόνισε ο συνάδελφο Άντεχ. Έχετε δίκιο, διότι όντω διαπράχθηκε ένα σφάλμα και σήμερα δεν είμαστε υπερήφανοι, δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την οδηγία αυτή μια οδηγία που δεν θα μας επέτρεπε να έχουμε τη δυνατότητα μαγνητικού τομογράφου. Όμως προσέξτε διότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ περιορισμένος και δεν μιλώ για τη σημαίνη μας συνεδρίαση, μιλώ για το χρόνο εφαρμογής της οδηγίας του 2004. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2012. Πρέπει λοιπόν να βρούμε όλοι μαζί τη διέξοδο για αυτό το κείμενο του 2012, ούτως ώστε να έχουμε μια απόλυτα ισορροπημένη λύση ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων, που είναι το βασικό θέμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε εμείς στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αφενός και της χρήσης της μαγνητικής τομογραφίας αφετέρου, την οποία χρειαζόμαστε για διαγνωστικούς σκοπούς, για την έρευνα, ε, για μελέτες ε, και απολογιστές σχετικές μελέτες γιατί η μαγνητική τομογραφία, όπως έλεγε ο Φιλίπ Ζουιβά, που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, είναι μια μέθοδος που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη τεχνολογία. Θα χάναμε λοιπόν ένα μέσο πολύτιμο για διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουμε οργανώσει μια ομάδα με όλους τους σκιώδεις συζήτητες, ούτως ώστε να μπορούμε όλοι να έχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για αυτό το πολύπλοκο θέμα και να μην, να μην μας διαφύγει τίποτα. Επίσης, δύο φορές κάναμε διαβούλευση με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα και με εκπροσώπους προσωπικού, γιατί είμαι ε, πρόεδρος της ομάδας ε, ε, που συνεργάζεται με τις εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είχαμε πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε αυτές ε, τις συζητήσεις. Πρέπει να προσέξουμε το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο, διότι να μην ε, ξεχνάμε ότι στις 7 χώρες της, ε, που ανέφερε ο κύριος Άντερ, συμπεριλαμβάνεται και η Πολωνία. Και επειδή έχουμε Προεδρία της Πολωνίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην χάσουμε χρόνο γιατί μας πιέζει ο χρόνος για την οδηγία. Ελπίζω ότι όλοι θα καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες για να πείσουμε τους συναδέλφους να μην δεσμευτούμε τελικά από αυτή την αντική, την αναστέλουσα μειοψηφία. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Ζώζε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί δεν μπορώ να κάνω παραπάνω σχόλια. Καταλαβαίνω βέβαια πως όσοι πήραν το λόγο συμφωνούν απόλυτα με την εναλλακτική που επιλέγει αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλέον προβλήματα ε, για αυτούς τις τομογραφίες που είναι πολύ σημαντικές και που θα πρέπει να στηριχτούν, γιατί σκεφτήκαμε κι εμείς πως ε, η εναλλακτική που επιλέξαμε ήταν η καλύτερη, ε, πολύ καλά πλαισιωμένη και βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικέ εξαιρέσεις ε, για το στρατό, για παράδειγμα, και σε κάποιο βαθμό και για τη βιομηχανία. Όλες αυτές τις τοποθετήσαμε, δεν το συζητήσαμε σήμερα, είναι σημαντικές όμως, γιατί κάθε μία έχει τα δικά της ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Για να μην μακρηγορήσω, να πω πως με την τροπολογία 13 ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε γιατί έρχεται σε αντίφαση με το σύστημα της αναλογικότητας και ευελιξίας που προσπαθήσαμε να εισάγουμε στα παραρτήματα για να διευκολύνουμε την θέση σε εφαρμογή της οδηγίας και κυρίως ε, την αξιολόγηση του κινδύνου από τους εργοδότες. Το κείμενο μοιάζει πιο απλό αλλά δεν κολλάει με τη γενικότερη φιλοσοφία. Ένα τεχνικό θεματάκι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνω τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. 5 Δεκεμβρίου, τελική προθεσμία και στις 12 το μεσημέρι και στις 24 Ιανουαρίου θα το ψηφίσουμε και μετά στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αύριο στις 10 θα ξεκινήσει η ομάδα, 9 με 10 συντονιστές.